Good morning, uh, colleagues. Before we um, go to our... our... Καλημέρα, συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος. Πριν πάμε στο πρώτο μας θέμα που θα είναι το 13, όσον αφορά τα τον ΛΟΑΔ και τον κατάλογο των δράσεων, ούτως ώστε να α, υπάρχει περισσότερη ποιότητα. Στην οικονομική περισσότερη ισότητα για να δούμε τώρα Έχουμε πει, οπότε έχουμε αυτές τις ανακοινώσεις τώρα και κατόπιν να προχωρήσουμε όσον αφορά κάτι σημείς της και σήμερα το πρωί. Έχουμε το ψήφισμα ε, της Επιτροπής μας για τα δικαιώματα ε, των διαφυλιγών. Και οι συντονιστές ενέκλαν το κείμενο Σύμφωνα με το άρθρο 128, κατόπιν έχουμε τη γνωμοδότηση για τις έρευνες της Όλαφ και την ε, συνεργασία με τον Ευρωπαίο Ισαγγελέα Συμφώνησαν οι συντονιστές να υποβάλουν σε αγγλικά και γαλλικά τις ε, τροπολογίες. Τρίτον, η ΙΜΚΟ και η ΛΥΜΠΕ όσον αφορά τις αρμοδιότητές μας και τον κανονισμό για να μην υπάρχει διάδοση ε, της προπαγάνδας των τρομοκρατών στο ίντερνετ είπαμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 53 θα υπάρχει συναρμοδιότητα για το θέμα αυτό μεταξύ ημών και της ΙΜΚΟ. δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό, οπότε περιμένουμε. Επομένω, πάμε στο, στο άρθρο 53 συν όσον αφορά το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο ίντερνετ. Τέταρτον, Πολιτιστική Επιτροπή και ΛΥΜΠΕ και αρμοδιότητές μας έχουμε τον κανονισμό για πρόληψη του τρομοκρατικού περιεχομένου στο ίντερνετ. Οπότε οι συντονιστές είπαν θα πρέπει να απορριφθεί το αίτημα της Επιτροπής Πολιτισμού και ας γίνει γνωμοδότηση σύμφωνα είπαν με το άρθρο 53. Πέμπτο και τελευταίο. Έχουμε την ομάδα που εποπτεύει το τι γίνεται με την διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του κράτος δικαίου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για Μάλτα δηλαδή και Σλοβακία. Αυτή η ομάδα εργασίας, τέλος αυτή η εποπτική ομάδα, είπαν ότι θα, οι ότι θα ισχύσει η προθεσμία της 19ης Απριλίου για την ε, γνωμοδότηση. Θα πάμε στην ε, Ολομέλεια του Μαρτίου και πρόεδρος θα είναι η κυρία Νετφέλτ. Δεν θα χρησιμοποιηθεί ο κανένας ε, ντεόντ ή άλλος κανόνας για την κατανομή και στις 10 του θα ξαναζητεί ο θέμα στους συντονιστές. Συμφωνεί η Επιτροπή με αυτές τις προτάσεις των συντονιστών. Μάλιστα. Σας υπενθυμίζω ότι στις 9 και 4 θα γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Οπότε πάμε τώρα στο σημείο 13. Έχουμε την εβδομάδα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κοινοβούλιο και εδώ έχουμε την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΔ κατά πολέμηση δυσμενών διακρίσεων όσον αφορά τα θέματα ταυτότητας και σεξουαλικού προσανατολισμού. Στο Δεκέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αυτόν τον κατάλογο δράσεων και εμείς καλέσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει αυτόν τον κατάλογο δράσεων καθώς και το μελλοντικό πρόγραμμα εργασιών αυτό το σημαντικό θέμα. Οπότε να δώσουμε στον κύριο Σμιτ τώρα τον λόγο απλώς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατόπιν οι συνάδελφοι μπορούν να λάβουν το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας κύριε βουλευτές. Καταρχάς θα ήθελα να ε, σας ευχαριστήσω που δώσατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ευκαιρία να παρουσιάσει μια επικαιροποίηση για τον κατάλογο μέτρων της ε, ε, Κομισιόν για την πρόθεση των μέτρων ισότητας για τους ΛΟΑΜΔ. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα είναι η ε, Παγκόσμια ημέρα ε, μεσοφιλικών που λαμβάνει η χώρα στις 10 Νοεμβρίου κάθε χρόνο ε, για να θυμόμαστε ε, τους, να μνημονεύουμε τους ανθρώπους που δολοφονήθηκαν λόγω της εχθρότητας κατά των ε, μεσοφιλικών ανθρώπων. Ε, είναι μια μέρα ε, λοιπόν μνημόνευσης αυτών των ανθρώπων παγκοσμίω και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με αυτή την ευκαιρία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια ε, συγκριτική ανάλυση ε, για την ισότητα για τα μεσοφιλικά και διαφορικά, διαφιλικά άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτή Είναι μια εργασία όχι της, των υπηρεσιών της Κομισιόν αλλά ενός ανεξάρτητου σχετικά Υπάρχουν ιδιαίτερε ανάγκε αυτών των προσώπων, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει προς νομική προστασία, διότι ακόμη απόρο απέχουμε από αυτά που θα θέλαμε να γίνουν σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, θα ήθελα να σας τονίσω ότι στα περισσότερα από τα νέα κράτη-μέλη ακόμη δεν έχουμε ειδικέ διατάξεις για την προστασία αυτών των μεσοφιλικών. Για να επανέλθω στον κατάλογο των δράσεων, ε, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με, το προσ... με την πρόσφατη έρευνα του Ευρωπαϊκού Βαρομέτρου, 71% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν την άποψη ότι πιστεύουν ότι τα άτομα ΛΟΑΜ θα πρέπει να έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με οποιονδήποτε ετεροφιλόφιλο. Όμως, αν δούμε πώς ε, γίνεται αντιληπτή η κατάσταση και ποια είναι η εμπειρία των ίδιων των ατόμων ΛΟΑΜΔ, τότε βλέπουμε ότι σχεδόν το 50% των ατόμων αυτών, 45% συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι έχουν βιώσει διακριτική μεταχείριση ή παρενόχληση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Αυτό λοιπόν πραγματικά μας δείχνει ότι πολλά πρέπει να γίνουν. Και αν προσθέσουμε σε αυτό ε, τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και υπάρχει πεδίο για δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, ο κατάλογος των μέτρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά χρησιμοποιεί τις αρμοδιότητες της για την καταπολέμηση των διακρίσεων, αλλά ταυτόχρονα προσπαθεί να δίνει το καλό παράδειγμα και να εμπνέει τα κράτη-μέλη να αναλαμβάνουν δράση για να προωθήσουν ε, την ισότητα των ΛΟΑΜΔ. Όπως είπατε κύριε Πρόεδρε ήδη, το Δεκέμβριο του 2015 δημοσιεύσαμε τον κατάλογο των δράσεων που με ένα συνολικό τρόπο καλύπτουν όλους, όλους τους τομείς πολιτικής ε, που επηρεάζουν τους ανθρώπους ΛΟΑΜΔΑ. Μη διακριτική μεταχείριση, ε, εκπαίδευση, ε, υγεία, απασχόληση, ελεύθερη, ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, άσυλο και εξωτερική πολιτική. Η Κομισιόν τακτικά κάθε χρόνο ε, υποβάλλει αναφορά για τον κατάλογο των μέτρων με ε, ε, γραπτός. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω κάποια, να επισημάνω κάποια σημαντικά σημεία υπόψη των αξιότιμων κυρίων ευρωβουλευτών. Πρώτα απ' όλα ευαισθητοποίηση. Θεωρούμε ότι η ευαισθητοποίηση παραμένει ένας κρίσιμος παράγοντας για να ε, δείξουμε ότι υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει στο νομοθετικό επίπεδο, αλλά και απλώς ε, όσον αφορά την υλοποίηση των κανόνων στην καθημερινή ζωή. Γι' αυτό αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε βίντεο για όλα τα θέματα που αφορούν ε, τους αγώνες των ΛΟΑΜΔΑ, για τις ιδιαίτερες καταστάσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι άνθρωποι αυτοί και οι καταστάσεις αυτές παρουσιάζονται με ένα εύκολο, ευνόητο τρόπο για το ευρύ κοινό. Αυτά τα βίντεο ε, παρήχθησαν στην αρχή της χρονιάς βεβαίως, ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν ε, κατά την ε, ημέρα που είναι αφιερωμένη σε αυτά τα θέματα και στις ειδικέ εκδηλώσεις. Και φροντίσαμε ιδιαίτερο στα βίντεο αυτά να ε, διαχυθούν ε, ιδίω στα κράτη-μέλη όπου η κοινωνική αποδοχή των ΛΟΑΜΔ είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα διαφιλικά άτομα, όπως σας είπα, είναι ένα από τα θέματα που καλύπτουμε με τα βίντεο αυτά όπως ε, ε, αναφέρθηκε και ζητήσατε με ένα ψήφισμά σας και η Κομισιόν προσπαθεί να το κάνει. Πήγαμε όμως και πέραν αυτού, ε, δημιουργήσαμε ένα toolkit όπως λέγεται για τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών, ώστε ε, να μπορέσουν ε, ενεργά να συμμετάσχουν σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που οργανώθηκαν σε όλα τα κράτη-μέλη. Και οι περισσότερες αντιπροσωπείες όντως συμμετείχαν ενεργά. Πολλές από αυτές, παραδείγματο χάρη, σήκωσαν τη σημαία με το ουράνιο τόξο και επίσης ε, οργάνωσαν ειδικέ συζητήσεις σε μερικά κράτη-μέλη. Επίσης, πολύ σύντομα, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η υποστήριξη προς την κοινωνία των πολιτών είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο, ιδιαίτερα στις μέρες μας που συρρυκνώνεται ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή τη στιγμή Έχουμε 22 κράτη-μέλη όπου είναι ενεργό το πρόγραμμα RAC, όπως λέγεται, όπως είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Και ε, τελευταίο και εξίσου σημαντικό, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι με την τελευταία έκθεσή μας για την, τον κατάλογο μέτρων ενθαρρύνουμε το, τα κράτη-μέλη να κάνουν το ίδιο για αυτά που κάνουν τα κράτη-μέλη ε, στους ανάλογους τομείς. Και βλέπετε ότι στις εκθέσεις μας υπάρχουν αναφορές ε, και των κρατών μελών για το τι ενέργειες αναλαμβάνουν. Τώρα, ε, κατόπιν αυτού θα ήθελα να προχωρήσω παραπέρα και να σας πω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο ευρωβαρόμετρο το 2019 θέλουμε να ζητήσουμε, να ρωτήσουμε για δεύτερη φορά τους Ευρωπαίους πολίτες τη γνώμη τους για τα δικαιώματα των ΛΟΑΜΔΟ, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια σύγκριση. Μετά επίσης μπορώ να σας δηλώσω ότι ο Επίτροπος είναι πάρα πολύ ε, δεσμευμένος στην ε, επιτυχή ε, παράδοση του έργου αυτού ε, στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τις πολιτικές αυτές. Σχεδιάζει λοιπόν να οργανώσει μία εκδήλωση προς το τέλος της θητείας αυτής της Επιτροπής, όπου να γίνει ένας απολογισμός για τα όσα θα έχουν επιτευχθεί μέσω του καταλόγου δράσεων και να εντοπιστούν τα περαιτέρω μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν. Και τέλος για να κλείσω, για να ολοκληρώσω την εικόνα, ζητήσαμε από τον Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για δεύτερη φορά να διεξαγάγει μια ε, δημοσκόπηση μεταξύ των ατόμων ΛΟΑΜΔ για το 2019, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τη σύγκριση από τις πληροφορίες αυτές, αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη στιγμή που αρχίσαμε αυτόν τον κατάλογο δράσεων και όταν θα ολοκληρωθούν το 2019. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ να μας ε, ε, ενημερώνετε τακτικά για τις εκδηλώσεις αυτές που θα λάβουν χώρα μέχρι το τέλος της θητείας. Και τώρα θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν σχόλια και να αναφέρω και ένα άλλο στοιχείο εδώ, το οποίο είναι το ψήφισμα, σχέδιο ψηφίσματος για τα δικαιώματα των ε, διαφυλικών ατόμων. Προετοιμάσαμε για το σκοπό αυτό ε, εν ώψη αυτής της συζήτησης ένα σχέδιο ψηφίσματος το οποίο βρίσκεται σε επίπεδο υπηρεσιών to the Commission and Council on the rights of intersex people pursuant to Rule 128. Ε, αυτά σύμφωνα με το άρθρο 182 έχετε ένα σχέδιο το κείμενο. Please um, look at this draft. Ε, οπότε κοιτάξτε για αυτό το σχέδιο εκεί που αναφέρει για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεσοφιλικών. Πρόκειται για κάποια θέματα που δεν τα γνωρίζει το κόσμος και κάποια θέματα πολιτικής για τα ζητήματα τα σχετικά με την παθολογικοποίηση ε, και τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων αυτών και των ανηλίκων μεσοφιλικών και ότι υπάρχουν δικές ανάγκες, χρειάζεται πλήρης ε, προστασία αυτού του δικαιώματο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. και τώρα οι συνάδελφοι μπορούν να σχολιάσουν τα αρχικά ε, όσα μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν ζητήσει διάφορες συνάδελφοι. Το λόγο με τη σειρά θα μιλήσει ο κύριο Κύρκος πρώτος. Κύριε Κύρκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τις δράσεις της Κομισιόν, θα σταθώ σημείο 7 για την πρόοδο εφαρμογή τους στα κράτη-μέλη και με λύπη βλέπουμε ότι η Ελλάδα, η χώρα μου, μένει πίσω σε μια σειρά από αυτές. Δεν στηρίζει τις ΜΚΟ για τις προκαταλήψεις κατά τον ΛΟΑΚΙ και μένει πίσω σε αυτές τις δράσεις που πολύ σωστά περιγράφει η Κομισιόν. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα, στις 21 Σεπτεμβρίου ένας νέος άνθρωπος κακοποιήθηκε ξυλοφορτώθηκε, λιντσαρίστηκε στο κέντρο της Αθήνας. Τα πρωτόγωνα αντανακλαστικά της κοινωνίας ξύπνησαν αμέσω. Ήταν ένα... Και η οικογένεια είχε να αντιμετωπίσει όχι μόνο τον πόνο για το χαμό του ανθρώπου, αλλά και τη δολοφονία του χαρακτήρα του. Ένα πρεζόνι το οποίο μπήκε για να κλέψει, τα ήθελε και τα άπαθε. Όμως ο Ζακ Κωστόπουλος δεν ήταν μόνος του, ενεργό μέλος της ΛΟΑΤ κοινότητας, με πλούσιο έργο, με πλούσια δράση, κινητοποιήθηκαν στη μνήμη του πια Δεκάδε σύλλογοι, οργανώσει, κόμματα, πολίτε, και έφτασε και μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Στι 25 Οκτωβρίου περί, το όνομά του ήταν μέσα στο ψήφισμα που βγάλαμε και ψηφίσαμε στο Στρασβούργο. Και το χειρότερο, χθε κυκλοφόρησε η έκθεση του Ιτριοδικαστή, η οποία διέψευδε ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών, ήταν καθαρό και δεν βρέθηκαν και αποτυπώματα πουθενά στο κατάστημα πάνω σε αντικείμενα. Δεν ήταν ένα τοξικομανής ο οποίο μπήκε να κλέψει που και αν ήταν πάλι έχουμε κράτο δικαίου, υποτίθεται ότι έχουμε. Ήταν ένα άνθρωπο ο οποίος υπέστη bullying και βρήκε την πρώτη πόρτα για να σωθεί και εκεί αντιμετώπισε την αυτοδικία και τελικά οδηγήθηκε στο θάνατο. Βλέπουμε λοιπόν πως έχουμε πολλά βήματα ακόμα να πορευθούμε σε αυτή την πορεία και χαίρομαι πολύ για όλα τα μέτρα που προτείνει η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Thank you. Sophie please. Η Σόφη Ινετφέλτ. Ε, ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εισαγωγή του και να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια αλλά και για την πιο δημόσια υποστήριξη της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα δικαιώματα των ΛΟΑΜΔ παραδείγματο χάρη ε, για την παρουσία της στις μεγάλες ε, ε, Pride Parades σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όμως θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα. Γιατί υπάρχουν μελέτες, καμπάνιες ενημέρωσης, υποστήριξη. Όλα αυτά βεβαίως είναι ευπρόσδεκτα. Αλλά θα ήθελα να ξέρω για να ρωτήσω γιατί δεν ε, λήφθησαν πρωτοβουλίε για νέα νομοθεσία. νομοθεσία. Παραδείγματο χάρη κάτι που ζητάει πολλά χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να ε, ε, εξισωθούν τα ομοφοβικά εγκλήματα με τα εγκλήματα ξενοφοβίας και ρασισμού. τι έχει κάνει η Κομισιόν για να προτείνει μια οριζόντια οδηγία κατά της διακριτικής μεταχείρισης που έχει κολλήσει, αν δεν κάνω λάθος, εδώ και 10 χρόνια. Επίση, τι γίνεται με την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας. Γιατί από ό,τι βλέπω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει απολύτω τίποτα κατά ε, της ε, λεγόμενης νομοθεσίας για την προπαγάνδα κατά των ε, γκέι που εφαρμόζεται σε ορισμένες χώρες όπως τη Λιθουανία. Και πρόσφατα υποβλήθηκε μια κοινοβουλευτική ερώτηση όπου ρωτούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι κάνει σχετικά με το common ruling όπως λέγεται ε, για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τι γίνεται για την επιβολή αυτού του κανόνα γιατί φαίνεται ότι ε, ε, ε υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν εφαρμόζουν αυτή την απόφαση του δικαστηρίου. Και τέλο, εντάξει, καλέ είναι όλε οι μελέτε κλπ. Αυτά είναι καλά και απαραίτητα. Αλλά θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι λίγο πιο θαραλέα και να παίρνει θέση σε πολιτικό επίπεδο. Φυσικά, μέσω ημών απευθύνομαι στους επιτρόπους, να παίρνουν θέση για θέματα όπως είναι ε, ισότητα στο γάμο. Ε, σύντομα θα είμαστε στο 2019 και η Κομισιόν είναι τόσο επιφυλακτική στο να αγγίξει το θέμα αυτό ενώ πολλοί ε, γρήγορα ε, σπέβδει να πάρει θέσεις για τον προϋπολογισμό της Ιταλίας ή δεν ξέρω τι στο Ηνωμένο Βασίλειο ή άλλα θέματα. Αλλά εδώ πρόκειται για ένα θέμα που αφορά τις αξίες μας και υποτίθεται ότι αυτή η Κομισιόν είναι πολιτική Κομισιόν. Δείξτε τα χρώματά σας αγαπητέ, ε, αγαπητοί Επίτροποι. Και νομίζω ότι σε καταστάσεις όπως το πρόσφατο δημοψήφισμα στη Ρουμανία, όπου ευτυχώς απέτυχε, ε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 21ου αιώνα θα πρέπει να έχει το κουράγιο να υψώσει το ανάστημά τη για τις αξίες που υπάρχουν μέσα στις συνθήκες μας ε, για την ισότητα στο γάμο, παρόλο που δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι θέμα αξίας της Ευρωπαϊκής ε, ε Ένωσης. Θέμα αξιών. Thank you, Chair. And, um, I the... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα, ιδίω για την ε, ε, ημέρα που ε, μνημονεύουμε τους ανθρώπους αυτούς και τις αδικίες που έχουν υποστεί οι μεσοφιλικοί άνθρωποι. για το θέμα της ισότητας στο γάμο υπάρχουν όλες αυτές οι συμφωνίες ε, της ε, Μεγάλης Παρασκευής, υπάρχει το Brexit και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη Βόρεια Ιρλανδία ε, όπου τα προβλήματα για τους ανθρώπους ΛΟΑΜΔΕ συνεχίζονται επί δεκαετίες τώρα. Και όλα αυτά λόγω ενός πολιτικού το ίδιο που αρνείται το δικαίωμα στην άμβλωση, αρνείται και τα δικαιώματα των ανθρώπων ΛΟΑΜΔΑ στη Βόρεια Ιρλανδία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, γιατί υστερεί πολύ ε, το βόρειο κομμάτι της Ιρλανδίας. Μόνο 10% ε, ε, των εγκλημάτων που οφείλονται στους λόγους αυτούς αναφέρονται στην αστυνομία. ενώ είχαμε 472 τέτοια ε, περιστατικά. Και μόνο φέτος το πρόγραμμα για την παρακολούθηση ε, των προβλημάτων αυτών, TMM, αναφέρει 169 δολοφονίες ε, ανθρώπων με κάποια τέτοια διαφορετικότητα. Είναι πραγματικά σοκαριστικό και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντική αυτή η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων που γίνεται σήμερα. Ένας ε, στους τέσσερις ανθρώπους ΛΟΑΜΔΑ από την Βόρεια Ιρλανδία ε, προσπάθησαν να αυτοκτονήσουν τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους και ξέρω ότι και σε άλλες περιοχές αναφέρονται τέτοια νούμερα λόγω των διακρίσεων που υπάρχουν. Οι αριθμοί που, μαθαίνουν, που, παίρνουμε ε, και τα ποσοστά αναφοράς των εγκλημάτων αυτών στην αστυνομία, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά περιστατικά και ε, ποσοστά που δεν αναφέρονται στην αστυνομία σε όλα τα κράτη-μέλη, που δεν καταγγέλλονται. Ε, Υπάρχουν λοιπόν ε, κόμματα όπως το DUP και άλλα ομοφοβικά κόμματα στην ε, Βόρεια Ιρλανδία και είναι σοκαριστικό και απαράδεκτο ότι οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα αρνείται τα δικαιώματα ε, των ανθρώπων που αγαπούν ο ένας τον άλλον. Να μην μπορούν, παραδείγματος χάρη, να έχουν το δικαίωμα να παντρευτούν. Ε, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει πολύ περισσότερη δουλειά. Συμφωνώ με τα μέτρα που αναφέρει η Κομισιόν, αλλά τα βιώματα ε, που έχουν οι άνθρωποι αυτοί, η διακριτική μεταχείριση που αντιμετωπίζουν είναι πραγματικά κάτι το αβάσταχτο σε καθημερινή βάση και θα πρέπει οι ευρωβουλευτές να υψώνουν τη φωνή τους ε, για το θέμα αυτό και σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δώσετε να ανταλλάξουμε απόψη μας σήμερα και ελπίζω ότι η Κομισιόν θα κάνει πολύ περισσότερα πράγματα για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Έχουμε έναρξη των ψηφοφοριών στις 9 ε, και 4, μην ξεχνάτε. Θα παρακαλούσα να περιοριστείτε στο χρόνο σας, συνάδελφοι, παρόλο που το θέμα αυτό ξέρω ότι είναι πολύ ευαίσθητο. Κορνίλια. Κορνίλια, Ερνστ, Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πραγματικά και ευχαριστώ που βάλετε το θέμα στην ημερήσια διάταξη, γιατί πρέπει να γίνει θέμα και εδώ. Γνωρίζουμε ότι στις περισσότερες χώρες μέλη, αλλά βέβαια και εκτός από τις χώρε μέλη και σε άλλες χώρες, χωρίζονται τα φύλλα σε ανδρικό και θηλυκό, αρσενικό και θηλυκό δηλαδή. Αλλά υπάρχουν και άλλα. Και πρέπει να σπάσουν τα ταμπού. Αυτό δεν, σε αυτό δεν αρκούν μόνο νομοθεσίε. Χρειάζεται άλλου είδου παιδεία να αρχίσει από το σχολείο, αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι λάθο να θεωρεί κανεί ότι υπάρχουν μονάχα δυο φύλλα. Πρέπει να αντιληφθούν ότι για ανθρώπου πρόκειται. Μεγάλα προβλήματα έχουμε, αλλά και στη Γερμανία και αλλού, με την καταχώρηση στα Μητρώα, που θα γράφονται οι άνθρωποι δηλαδή. Σε άλλε χώρε βέβαια τα πράγματα είναι πραγματικά πολύ χειρότερα. Στη Γερμανία ε, ακόμα θεωρούν ορισμένοι ότι πρόκειται για αρρώστια, δηλαδή κάτι το οποίο ξεφεύγει από το κανονικό. Ακόμα και χειρουργικές επεμβάσεις κάνουν σε πολλές χώρες για να διορθώσουν, να επαναφέρουν στην τάξη των εισαγωγικών φυσικά. Και η αυτοδιάθεση, ο κάθε άνθρωπος δηλαδή να αποφασίζει για το σώμα του, αυτό το καταστρέφουν, για να μην μιλήσω για τις πράξεις βίας. Το θέμα είναι σημαντικό. Χρειαζόμαστε νομοθετικά μέτρα, χρειαζόμαστε όμως και πάρα, πάρα πολλή δουλειά δημοσιότητας. Ελπίζω να μην ξαναγίνει αυτό, δηλαδή να έρθουμε εδώ 8.30 ώρα το πρωί για να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Πρέπει να γίνει θέμα, μέγα θέμα και να συζητηθεί. Αν δεν μπορεί ο άνθρωπος να αποφασίσει ποιο είναι, τι είναι και πώς ζει, όλα τα υπόλοιπα είναι περιτά. Όταν τελικά ο ίδιος ο άνθρωπος δεν ξέρει τι είναι ή τι του επιτρέπεται να είναι. Είναι μέγα θέμα λοιπόν αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε και πρέπει να παραμείνουμε, να επιμείνουμε, να εμείνουμε στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Κορονιλία. και ευχαριστώ που πραγματικά τα είπε συνοπτικά και έμεινε μέσα στα χρονικά όρια. Ακολουθεί Julie Ward. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που ε, φιλοξενούμε αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση. Δεν είμαι μέλος της ΛΥΜΠΕ, είμαι της, ομα... της ΦΕΜ, αλλά βρίσκομαι εδώ γιατί στην Επιτροπή ΦΕΜ μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα θέματα αυτά και των γυναικών και το, της κοινότητας του ΛΟΑΜΔΙ και θέλουμε να εργαζόμαστε ε, για όλα αυτά τα θέματα μαζί. Ε, στην παρουσίαση ε, Παρατήρησα τη διαφορά ανάμεσα στο πώς αντιλαμβάνεται το θέμα ε, το ευρύτερο κοινό και πώς ε, η ίδια η κοινότητα ΛΟΑΜΔΟ όσον αφορά ε, τα δικαιώματά τους. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει το χάσμα που υπάρχει λόγω της δομής των εξουσιών που έχουμε και την κυριαρχία των ανδρών στα εκλεγμένα σώματα, την έλλειψη εκπροσώπησης των ΛΟΑΜΔ. Αυτό σημαίνει ότι ε, δεν αισθάνονται ε, ε, οι άνθρωποι αυτοί άνετα γενικότερα στην κοινωνία. Αισθάνονται ότι δεν τις ακούγονται από αυτούς που έχουν την εξουσία, ότι δεν τους παίρνουν στα σοβαρά. Πρέπει να το διευκολύνουμε λοιπόν, να, να διευκολύνουμε την ε, ε, ενσωμάτωση τους, να τους ε, παροτρύνουμε, να τους ενθαρρύνουμε, να ε, τους διευκολύνουμε να πάρουν θέσεις εξουσίας. Ε, ανησυχώ για τα θέματα αυτά, για τα δικαιώματα των Λάμδα σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit, γιατί η συνάδελφος αναφέρθηκε στο πρόβλημα της Βόρειας Ιρλανδίας. Βέβαια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τέλεια τα πράγματα, αλλά ο χάρτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τουλάχιστον παρέχει ένα δίκτυο ασφαλείας για τις μειονότητες. Ε, παρατηρώ ανθρώπους που παίρνουν θέσεις εξουσίας ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο για να εφαρμόσουν το Brexit και κάποιοι από αυτούς πραγματικά είναι ομοφοβικοί. Η Τερέζα Μέη λέει ότι θα απαλλαγεί από το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και βάζει σε θέσεις εξουσίας άνθρωποι που πραγματικά είναι κατάλληλοι για την ε, ε, υπεράσπιση αυτών των δικαιωμάτων. Έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα λοιπόν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και τέλος ήθελα να πω ότι το Σαββατοκυριακό ήμουν στην Ουκρανία όπου συνεργάστηκα με βουλευτές ε, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΜΔΑ ε, και άλλων στην Ουκρανία. Ε, Πρέπει να ε, σας πω ότι σχετικά με τις χώρες αυτές που βρίσκονται καθοδόν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει εμείς οι ίδιοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να ε, έχουμε καλύτερες επιδόσεις. Χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα για να ενθαρρύνουμε και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα αυτά των ανθρώπων και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριο Γιούρεκ, παρακαλώ, προσπαθήστε να μείνετε μέσα στα δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μιλείτε για ανθρώπινα δικαιώματα διαφόρων ανθρώπων, για την αξιοπρέπεια. Βεβαίως, δεν υπάρχει θέμα ότι αυτό πρέπει να είναι ο κανόνας και είμαστε υποχρεωμένοι να τα σεβόμαστε τα πράγματα αυτά. Δεν είναι κάτι τα οποία μπορούμε να αποφασίσουμε εδώ να τα συζητήσουμε και να αποφασίσουμε ναι ή όχι. Όμως η κοινωνική διάσταση είναι κάτι που μπορεί και πρέπει να συζητηθεί. Και σε αυτή τη συζήτηση ακούμε συχνά να μιλούν για ισότητα στην κοινωνία. Θέλετε δηλαδή να βάλετε το σημείο της εξίσωσης ανάμεσα σε έναν άντρα και μια γυναίκα και για το γάμο και να επιτραπούν γάμοι ομοφύλων. Για μας όμως ο γάμος είναι ένωση ανδρός και γυναικός που από την ένωση αυτή μπορεί να προκύψει ζωή. Όταν μιλείτε για κοινωνικές νόρμες και έχουμε τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, εκεί ο ορισμός του γάμου είναι γραμμένος στα συντάγματα. Κάναμε και δημοψήφισμα στη Σλοβενία και στην Κροατία και οι άνθρωποι μαζικά τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης του ορισμού αυτού και του συνταγματικού αυτού ορισμού. Βεβαίω έγινε και δημοψήφισμα στη Ρουμανία που δεν ήταν νομικά δεσμευτικό. Σύμφωνοι. Αλλά πρέπει να ενδιαφερθούμε και για το τι λέει η πλειοψηφία. Υπήρξε σαφής πλειοψηφία υπέρ της διατήρησης αυτών των παραδοσιακών αξιών. Εφόσον θέλουμε να είμαστε δημοκρατικοί και να λεγόμαστε δημοκρατικοί και δημοκράτες, οφείλουμε να ακούσουμε και αυτές τις φωνές. Όταν θέλουμε να υπερασπιστούμε τη μονογαμική οικογένεια, αυτό δεν το πράττουμε κατά κάποιου άλλου ενάντια σε κάποιον άλλον. Το κάνουμε για να εξασφαλίσουμε το μέλλον τη Ευρώπη, και θέλουμε και εμείς να γινόμαστε σεβαστοί. Όταν ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας, είπατε, μας είπαν ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τις αξίες μας αυτές και εμείς θέλουμε να γίνονται σεβαστέ. Μάρλιν Μπιόρκ. Ακούσαμε ένα από τα παραδείγματα μόλις τώρα φωνών της πλειοψηφίας που λένε ότι έχουν το δημοκρατικό δικαίωμα να δυσδύουν, να βάζουν χέρι στα δικαιώματα των μειονοτήτων. Είπε πολλά για αξίες και τι αποφασίζουμε ως ελάχιστο δημοκρατικό σύστημα. Όμως εκεί χορηγούνται δικαιώματα στις μειονότητες. Και μάλιστα μόλις εγκρίναμε και γνωμοδότηση. Δέχομαι και χαιρετίζω το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία δίνει τα δικαιώματα να ζω όπως θέλω με την οικογένειά μου. Είναι ανισχυτικό, αλλά εν πάση περιπτώσει το αναγνωρίζω. Τώρα, είναι σημαντικό να δούμε ότι σε ορισμένες χώρες έχουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις, όπως Πολωνία, Ουγγαρία, Λιθουανία, αλλά και σε άλλες, και σε άλλες χώρες, όπου παραβιάζονται τα δικαιώματά μας. Σε άλλες χώρες τα πράγματα πάνε σωστά και αυτό πρέπει να το δούμε και να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο αυτή την κίνηση. Είναι καθαρό για μένα ότι η ομοφοβία και η τρανσφοβία που βλέπουμε συνδέονται με δεξιούς εθνικιστικούς, μάλλον εθνικιστικές κινήσεις και πρέπει να δράσουμε κατά των δυνάμεων αυτών. Και μάλιστα διακομματικά, υπερκομματικά. Ήθελα να πω και άλλα πράγματα, αλλά θα επαναλάβω αυτό που είπε η Σοφίντ Φέλτ για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν κάνει. Μιλούμε για εγκλήματα μίσους Μιλούμε για την ελευθερία της διακίνησης, της κυκλοφορίας και το νόμο προπαγάνδας που έχει εγκριθεί στη Λιθουανία. Εγώ έχω να προσθέσω το εξής. Είναι Trans Remembrance Day σήμερα. Έχουμε πολλούς, πολλές χώρες ακόμα όπου άνθρωποι ε, διεμφυλικοί ακροτηριάζονται για να επανέλθουν στην όρμα. Και αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη του 2018. Και κάτι άλλο που θέλω να τονίσω. Και θα τονίσω το ίδιο όταν θα έρθει και ο επίτροπο. Ότι το κράτο δικαίου συνδέεται με τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και με τα δικαιώματα των LGBT. Και αυτό που βλέπουμε στην Πολωνία είναι ότι το σύστημα δικαιοσύνη δεν είναι πλέον ανεξάρτητο. Και βλέπουμε πώ παρεμβαίνουν από το πολιτικό επίπεδο στην δικαιοσύνη και για θέματα LGBT. Θέλω να δω περισσότερη χρηματοδότηση και όταν μιλούμε για χρηματοδότηση, μη λησμονείτε το λάμδα, το L, τις λεσβίες. Και γίνεται και διάσκεψη κορυφής στην ε, Λιθουανία, το, την Άνοιξη. Και πολλές από εμά θα είμαστε αλλού απασχολημένες. Αλλά να πάτε όσους και όσοι μπορείτε εκεί. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ένα λεπτό, αλλά πραγματικά ένα λεπτό, Φερνάντο. Και μετά συνοψίζουμε. Θα είμαι πολύ σύντομος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωτών Δικαιωμάτων των Ευρωπαίων Πολιτών είναι χάρτης της τελευταίας γενιάς. Στο άρθρο του 9 λέει ότι ο γάμος είναι ένωση δύο προσώπων και προστατεύεται από τον νόμο, χωρίς καμιά διάκριση φύλου των μελών του, του δεσμού αυτού. Αυτό είναι ευρωπαϊκός νόμος. Δεύτερο, υπάρχει υπόθεση ότι ο ευρωπαϊκός νόμος, το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν αναγκάζει τις χώρες μέλη να νομοθετήσουν υπέρ γάμου ομοφύλων. Όμως, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η αμοιβαία αναγνώριση λειτουργεί έτσι ώστε καμία χώρα μέλο δεν θα πρέπει να προβάλλει ένσταση στην ελεύθερη κυκλοφορία εγκάμων ομοφύλων και ανθρώπων οι οποίοι έχουν αλλάξει το φύλλο τους. Στο ε, Μητρό... στο ληξιαρχείο. Και Αυτά ισχύουν ως νόμος. Ο ορίζον τον οποίο βλέπω είναι συνταγματική δημοκρατία καλή ποιότητα, όπου τα δικαιώματα του ατόμου δεν εξαρτώνται από την πλειοψηφία ούτε από τα αποτελέσματα δημοψηφισμάτων. Η δημοκρατία ποτέ δεν υπήρξε ο κανόνας της πλειοψηφίας. Αλλά κανόνας της πλειοψηφίας με σεβασμό της μειοψηφίας και με θεμελιώδη δικαιώματα και θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι ομόφυλοι, οι οποίοι είναι ελεύθεροι και επιθυμούν να δημιουργήσουν μια ένωση αστικού δικαίου, αλλά και γάμο με άλλον του ιδίου φίλου. Άλλο άτομο δηλαδή του ιδίου φίλου. Ευχαριστώ. Επιθυμώ να ευχαριστήσω ε, τα μέλη μας για τις ε, της υψηλής παρεμβάσεις, πρωί-πρωί κιόλας, αλλά είναι πολύ σημαντικό που κάναμε τη συζήτηση αυτή, διότι έχουμε σχέδιο ψηφίσματος και προφορική ερώτηση για ένα πολύ ευαίσθητο ε, θέμα τη σημερινή ημέρα δηλαδή. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, παρέμβασή της. Δεν προλαβαίνουμε τώρα να σας δώσουμε ξανά το λόγο. Πολλές από τις ερωτήσεις που ε, έθεσε η Σοφίν Φέλτ αλλά και άλλοι για την οριζόντια οδηγία, θα έχουμε βέβαια κάποιο χρόνο ίσως πριν από το τέλος ε, της κοινοβουλευτικής θητείας για να επανέλθουμε στις ερωτήσεις αυτές. Σας παρακαλώ σημειώστε τες εσείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις ε, ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών γιατί ήταν και θέματα ουσιώδη και θα τα ξαναδούμε για το ψήφισμα. Ευχαριστώ πολύ. Αντιλαμβάνεστε ότι ε, πρέπει να προετοιμαστούμε τώρα για την ψηφοφορία που αρχίζει σε περίπου ένα λεπτό. Colleagues, if everyone's ready, we can begin the votes. Αν είστε έτοιμοι συνάδελφοι, μπορούμε να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Μόνικα, ξέρω ότι εσείς είστε έτοιμοι. Μιλάω για όλους τους άλλους. Συνάδελφοι, πάμε τώρα στο 15 που είναι η πρώτη ψηφοφορία για τις κοινωτικές στατιστικές, για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία. Um, the, um, the is Cecilia Wickstrom. Η συγκεκριά είναι η Σεσίλια Βίξτρομ. Σεσίλια, θέλει ε, τον λόγο πριν ψηφορία. Ωραία, τότε προχωρούμε. Ψηφίζουμε με την τροπολογία 56. Vote is closed. Πέρα ψηφορίας. Ψήφισαν όλοι. Ωραία. Απορρίπτεται. 58 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 57. Πέρας. Συγγνώμη, συνάδελφε. Αυτό ήταν λάθος. Συμβαστική 1. Ψηφίζουμε. Θέλει προσοχή. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Ψηφίζουμε. 62. δύο. Συμπαθάτε με συνάδελφε, Πάμε στο 62. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 63. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 64. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Σελίδα 15 στο δικό μου κείμενο ψηφίζουμε. Συμβαστική 3. Ξαναλέω πρόεδρος, πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Ψηφίζουμε. Δεκαέξι, λέει γραμματείας, πέρας. Compromise Συμβαστική 5. Ψηφίζουμε. The vote is closed. Πέρα ψηφοφορία. Και εγκρίνεται. 148. 22. Σελίδα 22. 148. 148. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 149. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται αιτιολογίες παράγραφα. Τροπολογία 37. Ψηφίζουμε. Πέρας. 38. Εγκρίθηκε 37. Πέρας. Εγκρίνεται. 39 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 40 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 41. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 42. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 43. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 44. Πέρασε ο εγκρίνεται. 45 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 46 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 47 ψηφίζουμε. Πέρας, Απορρίπτεται. 48 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 49. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 50. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 51. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 54 ψηφίζουν. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ονομαστική. Πέρασε. Εγκρίνεται. 36, 4 χωρίς αποχές. και τελική ψηφοφορία για απόλυτη πλειοψηφία. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 36, 4 με 1 αποχή. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια, Ευχαριστώ. Η επόμενη ψηφοφορία είναι η γνωμοδότηση για θέσπιση στο πλαίσιο του Ταμείου Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συνόρων Μέσου Στήριξη. Είναι της ΙΜΚΟ. Γερούν Λέναρτς είναι ο εισηγητής. Γερούν, θέλεις το λόγο. Δεν είναι εδώ, άρα πώς θα μιλήσει. Πάμε στην ψηφορία. Τροπολογία 16. Ψηφίζουμε. Πέρασε ο φορέας. Εγκρίνεται 17. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 18. Ψηφίζουμε. You just thought you'd just interrupt me randomly. Okay, thank you. The vote is closed. And that's rejected. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 3. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 4. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 19. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 20. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Ψηφίζουμε. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22. Ψηφίζουμε. Closed. Πέρασε. Απορρίπτεται. 23. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Και εγκρίνεται. Η αιτιολογική 7. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 8. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 9. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 10. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 11. Ψηφίζουμε. Πέρας. απορρίπτεται 12 ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται 13 13 ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται 1 ψηφίζουμε Πέρας. Εγκρίνεται. 14. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 15. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τελική ονομαστική ψηφοφορία. ψηφοφορία 37, 1 με 4 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και πάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία για τις κοινέ διατάξεις όσον αφορά αυτό το Ταμείο για Οικονομική Στήριξη για τον Εξοπλισμό, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συνόρων, Ελέγχων κλπ. Ψηφίζουμε. Συμβαστική 11. Ψηφίζουμε. Πέρας. Θα πρέπει να αναφέρω τον εισηγητή που είναι ο Τόμας Σντεχόφσκι. Εγκρίνεται. 16. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Το 112 το, ή το 12 λέει τώρα ο πρόεδρος ε, έχει καταπέσει, συγγνώμη. 16 ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 84 ψηφίζουμε. Vote is closed. Εγκρίνεται συμβαστική. Ένα ψηφίζουμε. ο φορείος. Εγκρίνεται 95. Ψηφίζουμε. Ενενήντα πέντε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 2α, συμβαστική 2α. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 2β. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 96. Ψηφίζουμε. Πέρασε. κρίνεται. 105 ψηφίζουμε. Closed. Πέρα ψηφορίας. Amendment 106. Vote is open. 106. Ψηφίζουμε. Closed. Carried. 107. Εγκρίνεται. 107. Ψηφίζουμε πέρας και εγκρίνεται 108 πέρας εγκρίνεται 20 ψηφίζουμε πέρας εφορίας εγκρίνεται 109 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 110. Ψηφίζουν. Πέρασε. Εγκρίνεται. 21. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 22. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 111. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 23. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 113. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 114. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 115. Ψηφίζουν. Closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Closed. That's carried. Πέρας και εγκρίνεται. 118. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται 120. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 121. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 28. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 4α. Συμβιβαστική. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 4β. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται και αυτή. 127. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 128. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 129. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 130. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 131. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 132. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 133. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 134. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 135. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 136. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 137. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 32. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 33. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 138. Ψηφίζουμε Πέρασε. Απορρίπτεται 139. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται 134. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται 141 και 142 που είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται 143. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται 144. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται 145. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 34 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 146. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 148. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Πέρασε. 149 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 153 ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 154. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται 155. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται 156. Πέρασε. Εγκρίνεται 157. Πέρασε. Εγκρίνεται 158. Πέρασε. Εγκρίνεται 159. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται 160. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται 161. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Ψηφοφορία αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 177. Τροπολογία 177. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 178. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. απερίφθη. Συμβαστική 9 αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 181 αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 183 αρχίζει. Πέρας εγκρίνεται. 184 αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 185 αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Και αυτή η συμβαστική 10 αρχίζει. Πέρας εγκρίνεται. 189 αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 190 αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 191 αρχίζει. Πέρας απορρίπτεται 192 αρχίζει πέρας εγκρίνεται 193 αρχίζει πέρας απορρίπτεται 194 αρχίζει πέρας εγκρίνεται 195 αρχίζει Πέρας. Εγκρίνεται. 196. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 197. Αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. 198. Αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. 199. Αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. 200. Αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. 202 αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. 201 αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. 203 αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. 204 αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. 205 αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα τα citations, τροπολογία 2. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Αρχίζει. Αρχίζει. Για την 3. Πέρας. Εγκρίνεται. 44. Ε, στα recitals, δηλαδή στις αιτιολογικές σκέψεις. Πέρας. Απορρίπτεται. 45. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάντα σε αιτιολογικές σκέψεις, τροπολογία 5. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 47. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Την ψήφισαν 47. Συμβαστική 14 αρχίζει, συγγνώμη, αρχίζει η ψηφοφορία. 14 επαναλαμβάνουμε, επαναλαμβάνουμε την 14, γιατί την ψηφοφορία για την 14 δηλαδή, εγκρίνεται. 53 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. 44 άρχεται. Συγγνώμη, 54, 54. Πέρας. Εγκρίνεται. 50. 55 τώρα. 55, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 56, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. επτα Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15α. Άρχεται. Σε μένα λέτε Birgit. Ευχαριστώ, ναι. Ωραία, πέρας. Εγκρίνεται. 15β άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 9. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 60. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 61. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 62. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 63 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 64 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 11 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 13. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 14. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 67 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 68 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 69 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 70 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 71. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 72. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 73. Άρχεται.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 Απορρίπτεται. 77 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 78 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 79 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 80 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 81 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 82 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 83 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 15 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, ονομαστική αυτή, αρχίζει. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Πέρας. 31 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και 9 αποχές. Συγχαρητήρια στον Ισίδη. Τέλος της ώρας ψηφοφοριών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Okay, colleagues, we can resume our agenda um, if everyone is ready. Anyone who... Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να συνεχίσουμε αν είστε όλοι έτοιμοι. Όσοι δεν θέλουν να παρακολουθήσουν, να σβούν από την αίθουσα. Συνεχίζουμε με το σημείο 19, που είναι η ad hoc ε, αντιπροσωπεία τη Επιτροπή Λίμπε στη Σλοβακία και Μάλτα, 17 με 20 Σεπτεμβρίου του 2018. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η ad hoc αυτή αντιπροσωπεία στη Σλοβακία και τη Μάλτα είχε επικεφαλή στη Σόφι Ντεβέλτ ω πρόεδρο τη Ομάδα εργασία, και γενικά η εντολή ήταν να παρακολουθήσουν το θέμα της ε, διαφθοράς και της ε, ένομης τάξης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με έμφαση στη Σλοβακία και Μάλτα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Σοφή Εντεβέλτ για να μας παρουσιάσει την έκθεση από την αποστολή αυτή και μετά θα ακούσουμε τους σκιώδες εισηγητές και τους άλλους συναδέλφους για τα θέματα αυτά. Ε, Σόφη, θα ήθελες να μας παρουσιάσεις την έκθεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, λέει η κυρία Σόφια Εντεβέλτε. Ε, εκ μέρους της αντιπροσωπείας, με χαρά μου θα σας παρουσιάσω αυτή την έκθεση της αποστολής μας. Επισκεφτήκαμε την Σλοβακία και την Μάλτα σχεδόν πριν από δύο μήνες τώρα πια, 17 με 20 Σεπτεμβρίου και οι επισκέψεις αυτές ήταν η συνέχεια προηγούμενων ε, αποστολών μας, ε, της αντιπροσωπείας μας και στην Σλοβακία και στη Μάλτα. Βεβαίως όλα αυτά μετά από τη δολοφονία πρώτα της Δάφνης Γαρουάνα Καλίτσια και μετά του κυρίου Κούσιακ ε, που ήταν δημοσιογράφοι που ερευνούσαν διάφορες ε, ε, μορφές διαφθοράς, το οργανωμένο έγκλημα και ίσως σε σχέση με ε, τους πολιτικούς και ε, με την πολιτική. Ε, νομίζω ότι όλο αυτό το σημείο θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ε, στα πλαίσια αυτής της υπόθεσης. Λοιπόν, εξετάσαμε πρώτα απ' όλα τις έρευνες που γίνονται για τους δύο αυτούς φόνους και μετά γενικότερα την κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου σε αυτές τις δύο χώρες και τη λειτουργία των θεσμών. Ε, Έχουμε μία έκθεση που παρουσιάζει τα πραγματικά περιστατικά μας σε πολλές λεπτομέρειες, είναι 45 σελίδες και σε παράρτημα αναφέρουμε εξελίξεις που έχουν ε, μεσολαβήσει έκτοτε. Ε, για τις δύο αυτές έρευνες για τις ε, δολοφονίες καταρχάς και στις δύο περιπτώσεις οι δράστες οι ίδιοι έχουν συλληφθεί, αυτοί που διέπραξαν τις δολοφονίες. Στη Σλοβακία αυτό έγινε ε, πολύ γρήγορα μετά τη δική μας επίσκεψη και στις δύο περιπτώσεις όμως ε, αυτοί που βρίσκονται πίσω από αυτές τις δολοφονίες είναι ελεύθεροι. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσουμε ποια πρόοδος έχει γίνει στις έρευνες αυτές για τις ανθρωποκτονίες, γιατί για προφανείς λόγους η αστυνομία δεν μπορεί να μοιραστεί επιχειρησιακές λεπτομέρειες μαζί μας και αυτό είναι σωστό και δίκαιο, αλλά πρέπει να σας πω ότι παρατηρώ ένα διαφορετικό ύφο επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο αστυνομίες της ε, Μάλτας και της Σλοβακίας. Ιδιαίτερα ε, τις τελευταίες μέρες ε, στον τύπο υπάρχουν αναφορές που λένε ότι η αστυνομία της Μάλτας αναφέρει ότι έχει βρει τον εγκέφαλο ή τους εγκεφάλους που κρύβονται πίσω από τη δολοφονία της Δάφνης Καρουάνα Γκαλίσια αλλά είναι πολύ δύσκολο να ε, βρω τι είναι και τι δεν είναι αλήθεια γιατί αυτές είναι δηλώσεις στον τύπο, άτυπες δηλώσεις που στη συνέχεια διαψεύδονται, αλλά δυστυχώς αυτός είναι ο τρόπος ε, της επικοινωνίας και πρέπει να πω ότι είναι ευπρόσδεκτο ότι και στις δύο περιπτώσεις οι ε, δράστες, οι αυτούργοι τουλάχιστον έχουν ε, συλληφθεί και φαίνεται ότι αυτοί που συνελήφθησαν στη Σλοβακία είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με την αστυνομία και να δώσουν τις πληροφορίες που ξέρουν, ενώ αυτό φαίνεται να μην ισχύει στη Μάλτα. Ε, είναι όμως ε, υψηλής προτεραιότητας οι υποθέσεις αυτές. Ε, θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και ποτέ δεν θα πρέπει να περνάει ατιμόρυτη μια ανθρωποκτονία. Ε, με, γιατί έχει να κάνει με την ελευθερία και ασφάλεια των μέσων μαζικής επικοινωνίας, αλλά έχει να κάνει και με τους ε, ανθρώπους τους, ε, του, της οικογένειας των ε, θυμάτων. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία μόνο και όχι μόνο σε όλες τις λεπτομέρειες της έκθεσης αυτής. Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση και τα συμπεράσματά της. Αλλά θα ήθελα να αρχίσω με την Σλοβακία Έχουμε μία μεικτή εικόνα κάπως από τη χώρα αυτή. Υπάρχουν σαφώς ακόμα μεγάλες ανησυχίες, μεγάλα προβλήματα. Υπάρχει ακόμα ένα εχθρικό περιβάλλον για τους δημοσιογράφους και ο τελευταίος ε, Πρωθυπουργό Φίτσο ε, επισημαίνει ότι και πάλι έκανε κάποιε εχθρικέ παρατηρήσεις πρόσφατα εναντίον των ε, δημοσιογράφων και ελπίζω πραγματικά ότι οι σλοβακικέ αρχές θα λάβουν μια σαφή θέση εναντίον αυτού και θα δηλώσουν ότι θα διασφαλίσουν την ελευθερία και ασφάλεια των δημοσιογράφων όταν κάνουν τη δουλειά του. Υπάρχουν κάποια ανησυχητικά γεγονότα. Δεν ξέρουμε αν και σε ποιο βαθμό ερευνήθηκαν κάποια θέματα από τις αρχές. Παραδείγματο χάρη η περίεργη περίπτωση της απαγωγής ενός Βιετναμέζου ε, επιχειρηματία και ε, την επιθανή εμπλοκή του Υπουργού Εσωτερικών κυρίου Κάλινακ. Το θέμα της πύρας με τις μοτοσικλέτες επίσης ε, είναι ένα άλλο θέμα που έχουν και όπλα και τεθωρακισμένα οχήματα αλλά και πληροφορίες που προκύπτουν από τα Panama Papers, πληροφορίες που προσφέρθηκαν στις σλοβακικές αρχές από την γερμανική αστυνομία, αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα επίσης με τα ευρωπαϊκά ταμεία, ε, κονδύλια μάλλον για τη Γεωργία στη Σλοβακία. Ε, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει το γεγονός αυτό ε, τους ε, γεωργούς. Γιατί φαίνεται να έχουν εμπλακεί ανάμεσα στις ε, διαφορετικές αρχές. Βλέπουμε όμως και βελτιώσεις, σημεία βελτίωσης. Ε, γίνονται καλές προσπάθειες για να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο, παραδείγματο χάρη, διορίζεται ο αρχηγό της αστυνομίας ή οι δικαστές στο συνταγματικό δικαστήριο. Και παρόλο που δεν έχουν ληφθεί ε, ε, σχετικέ αποφάσει, βλέπουμε ότι γίνονται σοβαρέ προσπάθειες και ιδιαίτερα στην περίπτωση των ε, δικαστών, πριν από το Φεβρουάριο, 9 ναι, από τους 13 δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου πρέπει να αντικατασταθούν. Θα γίνει πολύ μεγάλος αριθμός λοιπόν διορισμών και σύμφωνα με τους νέους κανόνες θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και θα έχει επίσης και μεγαλύτερη επιρροή στο θέμα αυτό ο πρόεδρος. Ε, επίσης, ε, ε, ετοιμάζονται νέοι κανόνες για το διορισμό του αρχηγού της αστυνομίας. Η σλοβακική κυβέρνηση μόλις μας ενημέρωσε χθε με μια επιστολή για όλες τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει μετά από τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας αλλά και των Σέφερτς σχετικά με την ποιότητα της δικαστικής εξουσίας. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ ευπρόσδεκτα. Επίσης θέσαμε ερωτήσεις σχετικά με το RTVS, την ε, κρατική ραδιοτηλεόραση, ε, όπου ε, από ό,τι φαίνεται οι δημοσιογράφοι έπαιρναν οδηγίες σχετικά με το πώς να παρουσιάζουν θέματα που σχετίζονταν με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση όμως είπε ότι δεν έχει δώσει ποτέ επίσημες οδηγίες. Ένα συγκεκριμένο άτομο έδωσε κάποια στιγμή οδηγίες. Ε, αυτό ε, είναι κάτι το θετικό, αλλά παρόλα αυτά θα παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά ε, το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Θα παρακολουθούμε τις πιθανές θετικές εξελίξεις, αλλά θα ζητήσουμε και περαιτέρω μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και θα ε, παρακολουθούμε και το γεγονός ότι πολλά από τα μίντια βρίσκονται στα χέρια ολιγαρχών. Τώρα για την κατάσταση στη Μάλτα. Πρέπει να σας πω και αυτή είναι μια προσωπική μου παρατήρηση. Μας προβληματίζει βαθύτατα η κατάσταση στην ε, Μάλτα. Είναι δύσκολο να καταλήξουμε στο κατά πόσον υπάρχει κάποια έρευνα από πλευράς διοκτικών αρχών ή δικαστικών αρχών. Οποιαδήποτε έρευνα, από οποιονδήποτε και υπάρχουν καταγγελίες, υποψίες και θεωρούμε ότι θα πρέπει να ερευνηθεί εάν στέκουν οι σχετικές καταγγελίες, οι ισχυρισμοί, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο συμβαίνει κάτι τέτοιο. Από τις εφημερίδες, από τα μέσα ενημέρωση τα μαθαίνουμε. Σχετικά με την εταιρεία 17 Black που είχε κάποιες ε, ρυθμίσεις που τέλος πάντων πλήρωνε πολιτικούς και η ιδιοκτησία της ε, εταιρεία τώρα έχει εξακριβωθεί σε ποιον ανήκει και πρόκειται για ε, δύο μέρη της κυβέρνησης που τώρα είναι στόχοι ποινική έρευνας αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται έχει φτάσει η ώρα να παραιτηθούν αυτοί παραμένει εχθρικό το κλίμα για τους δημοσιογράφους, απειλούνται με μηνύσεις για συκοφαντία. Οπότε απευθύναμε έκκληση στην κυβέρνηση να εξασφαλίσει για το ότι αυτού του είδους εχθρική στάση κατά της οικογένειας της ε, Γκαρουάνα θα πρέπει να σταματήσει και το ίδιο να ισχύσει και για τις μηνύσεις επί συκοφαντία. Όμως δεν είμαστε σίγουροι ότι έγινε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση. Και υπάρχουν και κάποιοι που έχουν ανεγείρει ένα μνημείο για την Δάφνη Καρουάνα. Θα πρέπει τελικά να υπάρχει μια μεταχείριση ανθρώπινη. Πάντως, είναι θετικό ότι η κυβέρνηση της χώρας δέχτηκε την πρότασή μας να προσκαλέσει την Επιτροπή της Βενετίας ούτως ώστε να γίνει κάποιο είδου έλεγχο για το κράτος δικαίου, για τα θέματα των θεσμών, τα θεσμικά της ε, χώρας και αυτό θα γίνει μέσα Δεκεμβρίου. Γι' αυτό και ζητήσαμε να παραταθεί η προθεσμία όσον αφορά τη γνωμοδότηση, το, το πόρισμα της Επιτροπής ούτως ώστε να λάβουν υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας. Πάντως, εν κατακλείδη για τη Μάλτα προβληματίζομαι, ανησυχώ πολύ, πώς να το πω. Για το πόσα θέματα μας δημιουργούν προβληματισμό. Ξεβλήμα χρήματος, διαφθορά, απάτη, ενδεχομένως και παράνομη επιρροή των ψηφοφόρων, ε, τα όσα γίνονται σε βάρος των δημοσιογράφων. Πάρα πολλοί διορισμοί γίνονται έμεσα ή άμεσα από τον Πρωθυπουργό και το ιδιαίτερο γραφείο του. Μα πώς να γίνει η δουλειά με αμερόληπτο τρόπο από αυτούς. Όλα αυτά που μένουν είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Το τελευταίο μπορώ να σας πω αφορά τις χρυσές θεωρήσεις διαβατηρίων. Αυτό βέβαια δεν είναι αποκλειστικό ζήτημα ε, της ε, Μάλτας, γιατί υπάρχει διαφορετικό βαθμό σε πολλές χώρες και στη δική μου. Αυτή η πώληση, ας πούμε, διαβατηρίων. Η πώληση άδεια παραμονής ουσιαστικά είναι παράνομο εμπόριο τέτοιων ε, θεωρήσεων διαβατηρίων. Όλο αυτό είναι απειλή για το Σέγγεν ε, και για την ασφάλεια και για το κράτος δικαίου, για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας είπα, αυτό είναι προσωπική γνώμη, δεν το λέω ε, εξ ονόματος της Επιτροπής μας. Δεν νομίζω ότι αυτές οι τακτικές για τα διαβατήρια και τις βίζες είναι συμβατά και συνάδουν με τη συνθήκη του Σέγγεν. Δεν ξέρω να δούμε τι θα πει η Επιτροπή από πλευράς ε, των προτάσεων που θα διατυπώσει για τις χρυσές βίζες. Ξέρω ότι είχε αναλευθεί δράση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εποπτεία των τραπεζών και το ξέβλημα χρήματος. Θετικό και αυτό. Οπότε πρόεδρε, εν αυτά όσον αφορά τα βασικά σημεία της ε, έκθεσής μας. Και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ψήφισμα την άνοιξη του 19 σχετικά. Όπως ζητήσαμε, σας είπα αυτή την παράταση της προθεσμίας για να λάβουμε υπόψη τα συμπεράσματα της Επιτροπής της ε, Βενετίας. Στο μεταξύ θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε Μάλτα και Σλοβακία. ό,τι ό,τι ε, υποπέσει στην αντίληψή μα. οπουδήποτε. προ το παρόν όμω αυτέ τι δύο χώρε. Ο πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Τα μέλη τώρα τη ομάδα εργασία, αλλά και άλλοι συνάδελφοι μπορούν να λάβουν τον λόγο εφόσον το επιθυμούν. Έχω την Ρομπέρτα Μεζόλα, τον Ιώζεφ Βάιντεν Χόλζερ, την Κέμα Κοβέη και τον Σβέν Γκίγκολτ. Επιθυμεί άλλο, ο κ. Φρανς, άλλο, κανεί εξημών. Έχουμε χρόνο αν θέλετε να μιλήσετε. Καλώς. Κλείνω τώρα τον κατάλογο και η κυρία Μεζόλα, μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της ε, Ομάδας Εργασίας που πρόκειται, έχει για συζήτηση που παρακολουθείτε προσεκτικά και στην Μάλτα και στον Κόζο. Και είναι κρίμα που σε τέτοιο σημαντικό γεγονός δεν μπορώ καν να μιλήσω την μητρική μου γλώσσα. Ας το λάβει υπόψη η γραμματεία να υπάρχουν διερμηνείς δηλαδή για να μπορώ να μιλήσω τα μαλτέζικα. Ευχαριστώ πάντως την αντιπροσωπεία και ιδίως την Σοφίντ Φέλτ για την καλή δουλειά και τη συνεργασία την οποία είδαμε να αναβλύζει από όλο το φάσμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χρειάζεται δράση, χρειάζεται μια προσέγγιση βασισμένη σε πολιτική και τονίζει και πάλι την ανάγκη ενός μηχανισμού κράτους δικαίου που θα εξετάζει κάθε χώρα μέλος. Η αποστολή μας μας έδωσε μια ιδέα των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον, όταν θα, θα χρειαστεί διαφύλαξη του κράτους δικαίου σε όλες τις χώρες μέλη, με ε, διαφύλαξη της ελευθεροτυπίας και αγώνα κατά της διαφθοράς και της ατιμορρησίας. Τώρα πιο συγκεκριμένα για τη Μάλτα. 400 ημέρες έχουν περάσει από τότε που άνοιξε ο φάκελος του φόνου της, ε, μάλλον από τότε που έγινε η δολοφονία της Δάφνης Καρουάνα Γκαλίσια, η οποία τότε εργαζόταν πάνω σε μια πολύ σημαντική έρευνα κατά τη διαφθοράς και σε βάρος ε, μελών κυβερνήσεων και μάλιστα των ανώτατων ικριωμάτων τη κυβέρνηση. Στην έκθεσή μα περιλαμβάνονται ορισμένα σημαντικά συμπεράσματα μεταξύ αυτών και η ανάγκη να ενισχυθεί σημαντικά ο αγώνα κατά τη διαφθορά, καθώ και έκκληση προ τα πολιτικώ εκτεθειμένα πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση αυτή να διωχθούν. Μιλούμε και για τον νόμο κατά του ΣΛΑΠ, δηλαδή κατά της παρεμπόδισης των δημοσιογράφων ε, να ε, φέρουν τα θέματα ε, υπόψη του κοινού από ασυνείδητους πολιτικούς. Εδώ πρέπει να παίξει ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι δημοσίευση ενός stand-alone list που έχει αγοράσει εντό εισαγωγικών την ε, Μαλτέζικη ηθαγένεια είναι σημαντικό να γίνει διότι ξεπουλούνται τα Μαλτέζικα διαβατήρια και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Χρειάζεται να δημοσιευτεί η έκθεση πλήρως, διότι στην ολοκληρία της η έκθεση αυτή είναι γνωστή μόνο σε ορισμένα μέλη της κυβέρνησης. Και ο Υπουργό Κόναντ Μίτσι, που είναι ο μόνος ο οποίος εκτέθηκε από την υπόθεση των εγγράφων του Παναμά και ωστόσο εξακολουθεί να ασκεί εξουσία, αρνήθηκε να συναντήσει την αντιπροσωπεία και απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις για υποθέσεις μεταξύ αυτού και της ε, ε, επιχείρησης 70 Plus που βρίσκεται, έχει έδρα στο Ντουμπάι. Ζητήσαμε επίσης η εκστρατεία μίσους που ξεκινά συχνά από μέλη της κυβέρνησης κατά της οικογένειας και της μνήμης της Δάφνης Καρόνα Καλίτσια να πάυσει και να βρεθεί λύση για το αυτοσχέδιο μνημείο που ζητεί αποδομή δικαιοσύνη στην Βαλέτα. Είδαμε τις τελευταίες ημέρες ισχυρισμού ότι οι εγκέφαλοι πριν, πίσω συγγνώμη, από την ε, δολοφονία έχουν εντοπιστεί ή πάντως τους ακουμπούν. Δεν έχουν συλληφθεί ωστόσο, ούτε τους έχει ασκηθεί δίωξη. Η ε, λύση αυτού, η λυση αυτου εξυχνίαση αυτού του φόνου, αυτού του αποκρουστικού εγκλήματος είναι αναγκαία και για τη μνήμη της ε, ε Καρουάνα Γκαλίτσια αλλά και για τις υποθέσεις που διερευνούσε. Μέσα σε 400 ημέρες οι φωνές μας δεν έχουν μειωθεί σε ένταση ούτε και πρόκειται. Ευχαριστώ εκ μέρους Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ο Ιωσήφ Βάιντενχόλτσερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλα τα μέλη για την πολύ ε, έντονη δραστηριότητα. Το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει, υπάρχουν ακόμα πολλά ερωτηματικά για να ε, μάθουμε να αντιληφθούμε ποιος ανέθεσε ε, την εκτέλεση αυτών των φόνων. Αυτή είναι η κατάσταση για την ώρα. Δεν αποκλείεται να ζήσουμε εκπλήξεις στην υπόθεση αυτή στις επόμενες εβδομάδες. Ωστόσο, δεν μπορούμε να κρίνουμε ακόμη διότι δεν γνωρίζουμε ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις υποθέσεις, έστω και εάν ε, υπάρχουν κάποιες θεωρίες σχετικά. Είναι σημαντικό επίσης να δούμε πώς λειτουργούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είδαμε το έργο της Ευρωπόλ είδαμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε η εντολή διεξαγωγής ερευνών που έχει θεσπιστεί πρόσφατα. Η Ευρωπόλ υποστηρίζει και η προσπάθεια αυτή αποφέρει αποτελέσματα. Πρέπει να δούμε και πώς μπορεί να βελτιωθεί και το επιχειρησιακό έργο της Ευρωπόλ. Το ψήφισμα νομίζω πρέπει να περιλαμβάνει και αυτές τις πτυχές. Και στην Μάλτα αναμένουμε τα απορίσματα της Επιτροπής Βενετίας. η έκθεση της οποίας νομίζω θα δείξει εάν υπάρχει όντως συμβαστική παραβίαση του κράτους δικαίου στην Μάλτα. Συμφωνώ πάντως με την ιδέα και ψηφίσαμε άλλωστε στην τελευταία ολομέλεια στο Στρασβούργο ότι χρειαζόμαστε ανεξάρτητο μηχανισμό κράτους δικαίου για να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα αυτά σε πρώιμο στάδιο. Αυτοί οι δύο φόνοι μας έδειξαν πόσο σημαντική είναι η εμπλοκή του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με μια προσωπική παρατήρηση, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Ε, πιστεύω ότι πρέπει ε, να μπει η διαρεύνηση σε βάθος εις ό,τι αφορά την πώληση των ε, διαβατηρίων της Ιθαγένειας σε χώρες μέλη της Ένωσης, διότι αυτές είναι που ανοίγουν την πηξίδα της Πανδώρας. Εξεπλάγει που δεν είχαμε καν συνάντηση με αυτήν την εταιρεία που πολύ, ή οργανισμό, agency, λέει ο κ. Βάιντεν Χόλτσερ, που πολύ αυτές τις ηθαγένειες. Ευχαριστώ, Γιώζεφ. Κυρία Μακοβέη, είστε μέλος των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Αν θέλετε μπορείτε τώρα να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν θα μακρηγορήσω. Θέλω μόνο να πω ότι μετά από τις επανειλημμένες συχνές επισκέψεις στη Μάλτα και μία φορά στη Σλοβακία και τις συνομιλίες με τους απλούς ανθρώπους και τους ε, ε, επισήμους, δεν έχω καμία επιβεβαίωση ότι θα επιληθεί καμία από αυτές τις υποθέσεις. Και όταν μιλάω για επίλυση, διαλεύκανση, εννοώ να πιάσουν αυτούς που έδωσαν την εντολή. Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε τώρα στη Σλοβακία είναι οι δημοσιογράφοι είναι, ότι οι δημοσιογράφοι διαμαρτύρονται γιατί ένας ε, τέος ε, τους πρόσβαλε και πάλι και ότι πρέπει να παρουσιάζουν πληροφορίες για την χρηματοδότησή τους ε, και αποδείξεις, γιατί υπάρχει μια καταγγελία ότι χρηματοδοτούνται από τον Τζορτ Σόρος. Και ο ίδιος αυτός πρωθυπουργός ε, ε, ήταν αυτός που ε, βρισκόταν στην εξουσία όταν δολοφονήθηκαν ο Γιάννη και η σύντροφός του. Επίσης υπάρχουν πολλές αντιφάσεις στις δηλώσεις των επισήμων. Ε, και είναι περίεργο πώς ο καθένας ε, είπε διαφορετικά πράγματα για το τηλέφωνο που κατασχέθηκε ή για πολλά άλλα στοιχεία. Όσον αφορά τη Μάλτα, όπως είπε ήδη η Ρομπέρτα, ε, τίποτα δεν έχει αλλάξει πραγματικά. Και πάλι δεν περιμένω οι αρχές να φτάσουν αυτούς που έδωσαν την εντολή και μάλιστα υπάρχει ένα καινούριο σκάνδαλο που αφορά ε, ένα κονσόρτσιουμ συναδέλφων δημοσιογράφων της Δάφνης που αποκάλυψαν ότι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ε, πρόγραμμα ξεπλήματος χρήματος που αφορά 800 εκατομμύρια ευρώ και όπου εμπλέκονται ανώτατοι αξιωματούχοι της Μάλτας, ο Πρωθυπουργό, το Υπουργικό Συμβούλιο, ο κύριος Μίτσια κλπ. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από αυτούς τους ανθρώπους να ε, διεξαγάγουν έρευνες εναντίον του εαυτού τους. Αυτό θέλω να πω. Ελπίζω οι συνάδελφοι να βρουν την αλήθεια, αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι. Πρέπει να κάνουμε κάτι, γιατί αν οι αρχές δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, ε, η Europol ή κάποιος άλλος πρέπει να αναλάβει δράση. Δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι να ανακαλύψουν ποιος είναι ο δολοφόνος. Είναι πολύ θλιβερή η κατάσταση. Τώρα για την ε, αντιπροσωπή αυτή και την έκθεσή της δεν ξέρω πόσο βοηθάει. Βοηθάει να δείξουμε, ε, να γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά στην κοινή γνώμη, να δείξουμε ότι ενδιαφερόμαστε, ε, να πούμε ότι αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει και ότι οι έρευνες πρέπει να συνεχιστούν. Υπάρχουν εδώ παρόντα τρία μέλη της ομάδας εργασίας που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό, η κυρία Μόνικα Μπενόβα, πρώτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Μπένοβα. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ για την έκθεση. Για το σχέδιο του κειμένου όσον αφορά τη δήλωση. Είχαμε όλες αυτές τις ε, συναντήσεις, είχαμε ε, το ότι όπως γίνεται συνήθως δεν αναφέρεται το πλαίσιο στο οποίο έγιναν αυτές οι συναντήσεις. Συνεχώς προσπαθεί η κυβέρνηση να διεκπεριώσει τα εκκρεμή ζητήματα. Αυτό το επιβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός είχαμε οι ευρωβουλευτές μακρές συζητήσεις για τη γενική κατάσταση και για τα ζητήματα που αναφέρατε και είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε το ότι στη χώρα μας τηρούμε το κοινοτικό δίκαιο, σεβόμαστε τις δημοκρατικές αρχές πλήρως. Και θα πρέπει να σας τονίσω ότι αυτή η έκθεση πάσχει γιατί τα συμπεράσματα δεν αντικατοπτρίζουν κάποιες πλευρές αυτών των επαφών και συναντήσεων. Φερρυπίν δεν λέει για την συνάντηση με τον ειδικό εισαγγελέα όπου κατά λεπτός σας εξηγήθηκε το ότι το τηλέφωνο της κυρίας Χόλτσοβα κατεσχέθη και επεστράφη. Οπότε η έκθεση του Κοινοβουλίου δεν θα πρέπει να αφήνει να εννοηθεί το ότι υπάρχουν υποψίες που δεν είναι βάσιμες, που δεν υπάρχουν δηλαδή ε, κάποια επιβεβαιωμένα πραγματικά περιστατικά και να λέει εδώ ότι οι διοικητικές αρχές και άλλες αρχές έχουν επαφές με το οργανωμένο έγκλημα. Είναι επικίνδυνο στις εκθέσεις μας να λέμε τέτοια πράγματα όταν δεν υπάρχουν οι σχετικές αποδείξεις. Αυτά είναι απλές υποθέσεις, αβάσιμες. Είναι επικίνδυνο εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει τέτοια πράγματα στις εκθέσεις του. Η Σλοβακική κυβέρνηση ξέρει το ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα όσον αφορά την εμπιστοσύνη του κόσμου. Οπότε και θεσπίζονται αποτελεσματικά μέτρα κατά της διαφθοράς. για να υπάρχει επίσης περισσότερη ε, διαφάνεια όσον αφορά τους ε, διορισμούς, ιδίως όσον αφορά την αστυνομία. Τώρα όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι χωρίς ε, σύνορα θεωρούν ότι η Σλοβακία παίρνει πολύ καλό βαθμό στα σχετικά και ο κ. Κούτσακ δολοφονήθηκε αλλά δεν φταίει το ότι η νομοθεσία μας ε, είναι ανεπαρκής. 19 χρόνια είμαι πολιτικός και ανέκαθεν είχα πολύ καλές σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης και ο πρώην πρωθυπουργό, βέβαια ε, εκείνο είχε κάποιες προστριβές με δημοσιογράφους αλλά αν αυτό το θεωρήσετε ότι είναι μέτρια επίδοση της χώρας στα των ΜΜΕ είναι αβάσιμο. Δεν μπορείτε να το βάλετε αυτό στο κείμενο γιατί έχουμε, έχουμε ενδελεχή νομοθεσία και σε πολλά σημεία η δική μας νομοθεσία είναι καλύτερη από άλλων χωρών, πολλών άλλων χωρών. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε που ήρθατε στη Σλοβακία και που συναντήσατε εκπροσώπους της ε, κυβέρνησης, της ε, αστυνομίας, της δικαστικής εξουσίας, τους δημοσιογράφους και χαίρομαι για το ότι οι δημοσιογράφοι θέλουν να είναι αμερόληπτοι και αντικειμενικοί. Καλά, υπάρχουν κάποιες προστριβές με κάποιους πολιτικούς και κάποιους δημοσιογράφους. Και τονίζω το κάποιους. Ίσως θα ήταν γενικώ σωστό οι δημοσιογράφοι να έχουν καλύτερες σχέσεις με τους πολιτικούς και στα όσα ε, γράφουν να μην αποκαλούν τους πολιτικούς απατεώνες, κλέφτες και δολοφόνους. Μιλώ για κάποιους δημοσιογράφους, το αναφέρονται σε κάποιους από τους πολιτικούς μας. Ευχαριστώ. Okay, thank you. Um, uh, I'll the, the, um, the, uh, Ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Θα επανέλθουμε αργότερα στα θέματα αυτά. Κύριε Φραντς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να τονίσω την πτυχή της προστασίας των μειονοτήτων στην Σλοβακία. Η μεγαλύτερη μειονότητα στη Σλοβακία είναι άνθρωποι με ιστορικό Ρωμά που υφίστανται σημαντικότατο αποκλεισμό από το σύστημα παιδείας, από την στέγη και από την εργασία. Η κατάσταση αυτή που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί είναι εξαιρετικά αβέβαια. Πιέζονται για να καταλήψουν και τα αστικά κέντρα. Ακόμη και στην Ήπεθρο, όπου αναγκάζονται να κατοικούν, δεν υπάρχουν πάντοτε επαρκείς υποδομές και ταυτόχρονα υφίστανται εκμετάλλευση οι οποίοι αναγκάζονται να απασχολούνται με μισθούς πολύ κάτω των κατοτάτων. Πρόκειται για την πατρίδα των ανθρώπων αυτών ε, εδώ και 600-700 χρόνια και είναι υποχρεωμένοι να την εγκαταλείψουν διότι στη Σλοβακία ε, δεν έχουν πλέον ε, μέλλον, δεν έχουν δυνατότητα ύπαρξης. Ο αντιαθηγανισμός στην Σλοβακία και έχω μάλιστα πάει τρεις φορές εκεί πρόσφατα και μίλησα με τους ενδιαφερομένους οι οποίοι μου λένε ότι φτάνει πια ε, να παίρνει μορφή apartheid. Δεν ε, τους παίρνουν καν στα λεωφορεία ε, λόγω του ότι ανήκουν σε αυτή την ε, εθνική μειονότητα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να φωτίσουμε και δεν επιτρέπεται να το αφήσουμε να είναι ταμπού. Okay. okay. Okay. Okay, colleagues, okay. Ο πρόεδρος, ναι, ναι, σας, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Η κυρία Γκόμης. Ε, ευχαριστώ τις και τους συναδέλφους για την έκθεση της, ε, που καταθέτει η Σοφίν Τφέλτ καθώς και για τα σχόλια των συναδέλφων που συμμετείχαν. Ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα έγγραφα Παναμά που μετέβημε εκεί στη Μάλτα στα πλαίσια της υποθέσεως αυτής και ως επικεφαλής της ad hoc αποστολής για το κράτος δικαίου που μετέβη στην Μάλτα μέσω μετά την δολοφονία ε, εις βάρος της ε, Δάφνης Γαρουάνα Γαλήσια. Οφείλω να συμφωνήσω με τα όσα λέχθηκαν από την Σοφή Τφέλτ και από την Ροβέρτα Ματσόλα, Μετσόλα, συγγνώμη, ε, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της κατάστασης στην οποία προβαίνουν. Θέλω να τονίσω δύο πράγματα τώρα. Δύο απατεώνες, φοροφυγάδες, βεβαιωμένοι, διεφθαρμένοι, διευθύνουν το προσωπικό γραφείο του Πρωθυπουργού Σκέμπρη και πρώτα Υπουργό Ενέργεια, κ. Μίτσι, τώρα Υπουργό Τουρισμού. Τα άτομα αυτά εξακολουθούν να είναι μέλη τη Μαλτέζικη κυβέρνηση παρά το γεγονό ότι έχει καταδειχθεί όπως είχε γίνει και από την Ερευνητική Επιτροπή για τα Panama Papers, τώρα με τις πλέον πρόσφατες αποκαλύψεις για το Black 17 έχει καταδειχτεί ότι είναι απατεώνες, εγκληματίες. Και όμως είναι ακατανόητο πώς ακόμη αυτοί παραμένουν στην κυβέρνηση. Γιατί ο Πρωθυπουργό τους προστατεύει, γιατί δεν υφίστανται δίωξη από την ε, αστυνομία. Διότι διεξάγονται έρευνε από την μαλτεζική FIU, αλλά δεν τους απαγγέλει κατηγορίες η αστυνομία. Και υπάρχει και το μέγα ερώτημα σχετικά με την έρευνα για τον φόνο της Δάφνης Καρουάνα Γαλήσια. Όπως λέχθηκε προηγουμένως, βρίσκεται σε αδιέξοδο η έρευνα. Μάλιστα, συνελήφθησαν τρεις βομβιστέ. Το ερώτημα όμως είναι ποιος τους έδωσε τις οδηγίες, ποιος είναι ο εγκέφαλος ή οι εγκέφαλοι που δεν έχουν συλληφθεί. Και ορισμένοι ισχυρίζονται ότι κάποιοι θα πρέπει να ανακριθούν. Όμως ε, τα ίχνη αυτά δεν ακολουθούνται. Άλλωστε υπάρχει έκφραση μίσου και δαιμονοποίηση σε βάρος της οικογένειας της Δάφνης Καρουάνα με καταγγελίες περί, ε, με, μάλλον με δυσφημιστικές εκστρατείες με εξαίρεση έναν υπουργό που του ζητήθηκε να καταθέσει το ιστορικό των κλήσεων που έχει κάνει. Υπουργό Καντρώνα, Υπουργό Οικονομία, ο οποίο έπαυσε τι δυστημιστικέ εκστρατείε. Είπαν κάποιοι ότι τον είδαν να πίνει ποτά με κάποιον από του υπόπτου που έχουν φυλακιστεί ήδη ως ε, αυτούργοι της βομβιστική ενέργειας. υφίσταται διώξει αυτοί που ζητούν απονομή δικαιοσύνης και που έφτιαξαν το αυτοσχέδιο μνημείο. Και είναι απολύτως αποκρουστικό ο τρόπος με τον οποίο καλύπτεται το μνημείο και δεν επιτρέπεται στους ανθρώπους να αποδώσουν έτσι σεβασμό και τιμή στη μνήμη της Καρουάνα. Υπάρχει και μια δυσφημιστική εκστρατεία κατά των ευρωβουλευτών που ζητούν ενεργά υπονομή δικαιοσύνη, Ο συνάδελφο μα Ντάβιτ Κάσα, τον οποίο κατηγορούν για κατανάλωση ναρκωτικών και άλλα. Και πρόσφατα και για μένα την ίδια μου είπαν ότι βρέθηκα στην πρώτη γραμμή των ε, εφημερίδων που ε, επηρεάζει η κυβέρνηση και από ιστοσελίδες fake news σχετικά με την τελευταία μου επίσκεψη στο Καζακστάν στα πλαίσια αποστολής της Επιτροπής Εξωτερικών και λένε, διαδίδουν ότι έχω επαφές με τον Μουκτάρα Ζιαζόφ, με τον, οποίο έχω συναντήσει ποτέ. Πρόκειται για ιστοσελίδα που διακινεί fake news. Γράφουν και στην αστυνομία και, στην, ε, και στο Βέλγιο και στην Πορτογαλία. Και αυτό που βρίσκω ενδιαφέρον είναι ποιος κυκλοφορεί τα νέα αυτά, τα ψεύδια αυτά σε βάρος μου. Αυτοί όλοι είναι μέλη του κυβερνώντος κόμματος της Μάλτας και της Βουλής της Μάλτας. Είναι πράγματι αποκρουστικά αυτά που συμβαίνουν. Θυμούμε ότι τα ερωτήματα που θέσαμε σχετικά με το ξέβλημα χρήματος, ειδικά για την ε, τράπεζα Πιλάτος, αποδείχθηκαν αληθεί. Πρόσφατα άλλη τράπεζα έχει βρεθεί σε μεγάλους μπελάδες, μια Σάλτα Bank, τα ίδια, πλυντήριο βρώμικου χρήματος, εγκληματιών από άλλες χώρες. Βλέποντας τα όσα γίνονται, όχι μόνο στη Μάλτα, όπου υποσκάπτεται η δικαιοσύνη. Και αυτά που είπαν για την Σλοβακία. Θέλω να θυμίσω και την υπόθεση της Βουλγαρίας. Δεν δέχομαι ότι κάποιος τρελός δολοφόνησε και ιδίως διότι η Βικτόρια Μαρτίνοβα στη Βουλγαρία όπως ο Κουσάκ στην Σλοβακία και η Καρουάνα στη Μαλτά διερευνούσε υποθέσεις διαφθοράς και εξέθετε τους διεφθαρμένους. Και η βουλγαρική υπόθεση πρέπει να καλυφθεί λοιπόν από τι εργασίε της ομάδας εργασία Και μία ερώτηση προς την Σοφή. Η Ευρωπόλ κάποια στιγμή είπε σε επιστολή προς εμένα, την οποία έχω μάλιστα διανύμει, ότι η Ευρωπόλ αντιμετωπίζει περιορισμούς στην δράση της, ιδίως για τη Μάλτα. τονίζοντας ότι πρόκειται για κάτι παραπάνω, μια απλή δολοφονία, δηλαδή συνδέεται με εγκληματικές οργανώσεις. Και οι περιορισμοί ήταν το αποτέλεσμα ότι η εντολή τους δεν τους επιτρέπει να υπερβούν τα όρια που βάζουν οι αρχές. Μπορεί η Σοφίν Φέλτ να πει αν έχει έλθει σε επαφή με την Ευρωπόλ και αν έχει, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο, αν έχει ζητήσει και αυτή αυξημένη εντολή για την Ευρωπόλ για τις τρεις υποθέσεις. Μάλτα, Βουλγαρίας και Σλοβακία. Ευχαριστώ. Συναδελφοί, είχα κλείσει τον κατάλογο των ομιλητών, αλλά η κυρία Στύπερ και ο κύριο Νάτ ε, ήρθαν καθυστερημένοι. Αν γίνεται όμω να είστε πολύ σύντομοι, παρακαλώ. Ο κύριο Κρύπε πρώτα. Σας παρακαλώ όμω πολύ σύντομα και μετά θα δώσω το λόγο στη Σοφή για να απαντήσει στις ερωτήσεις που έγιναν. Ε, ο πρώτος ομιλητή για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι εύκολο σήμερα να μιλάει κανείς σε αυτή την Επιτροπή. Είμαι πεπισμένος ότι το κράτος δικαίου και οι σχετικές έρευνες δεν είναι το μίσο που θα πρέπει να επεμβαίνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι εσωτερικές υποθέσεις. Όμως μετά τη δολοφονία, η κατάσταση στη Σλοβακία, μετά τη δολοφονία του Γιάννα Κουσιάκ, Ε, λέω ότι μετά τη δολοφονία αυτή ε, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους. Αισθάνομαι όμως ότι πρέπει να μιλήσω υπέρ της Σλοβακίας ε, και ως μέλος αυτής της Επιτροπής. Ε, λυπάμαι πάρα πολύ που χρειάζεται να μιλάμε σήμερα τον 21ο αιώνα για τη δολοφονία δημοσιογράφων. Ο Γιάν Κούσιακ ε, έγραφε με πολύ ειλικρίνεια για εγκλήματα των πολιτικών, των αρχηγών της μαφίας και άλλων ε, εγκληματιών που υπάρχουν και δρούν στη χώρα μας. Μετά τη δολοφονία αυτή, πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν και οι δολοφόνοι του Κούσια και της Κούσνοβα ίσως δεν το περίμεναν αυτό. Περίμεναν ότι κάπως θα κουκουλωθούν αυτές οι δολοφονίες, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Ε, ε, ο κόσμος αντιδρά και πραγματικά είμαι πολύ απογοητευμένος που οι ε, αξιωματούχοι της κυβέρνησης μας δεν ε, πήραν τα ε, απαραίτητα μέτρα για να δείξουν την μια υπεύθυνη στάση. Ο κόσμος ζητάει δικαιοσύνη, αλλά βλέπουμε ο Πρωθυπουργό Φίτσο που εξακολουθεί να ζει σε ένα διαμέρισμα ε, που ε, ανήκει σε έναν φοροφυγά, ο οποίος καταδικάστηκε μάλιστα από τα δικαστηρία. Συγγνώμη, ε, αλλά είχε κλείσει ο κατάλογος, ο κύριος Νάτς πρέπει να μιλήσει στη συνέχεια. Τελειώστε παρακαλώ. Λοιπόν, πριν από μερικές μέρες ένας οπαδός του Κούσιακ είπε σε μια... Ε, ε, ο πατέρας του, συγγνώμη, είπε ότι αν όλοι κάνουν ε, σωστά τη δουλειά τους, ε, τα πράγματα θα πάνε καλά. Και αυτό από, τον, από έναν άνθρωπο που ο γιος του δολοφονήθηκε και απευθυνόταν προς τους πολιτικούς. Έχει λείψει η εντιμότητα και πρέπει να, ξα, να την ξαναβρούμε. Ευχαριστώ πολύ σύντομα ο κύριος Σνάτς. Ευχαριστώ. Δεν ήθελα να πάρω το λόγο, αλλά μετά από αυτά που ακούσαμε από τους συναδέλφους, ένα συνάδελφο μόλι έφυγε, ήταν ένα από αυτού, αλλά ήθελα παρόλα αυτά να πάρω το λόγο και να πω ότι στη Σλοβακία, ναι, έχουμε προβλήματα. Όπω παντού στην Ευρώπη υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν και αποκλεισμένε κοινωνικέ ομάδε. Όπω σε όλε τι ε, χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν προβλήματα με τι κοινότητε των Ρώμα. Αλλά σα παρακαλώ, εξ ονόματο τη Δημοκρατία τη Σλοβακία, σα παρακαλώ το ζήτημα δεν είναι ποιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Δεν υπάρχει apartheid, δεν υπάρχει αποκλεισμό των Ρωμά από τα δημόσια μέσα ε, συγκοινωνία στη Σλοβακία. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ε, δεν είναι πρόβλημα της σημερινής κυβέρνησης. Πολύ συχνά υπερβάλλουμε και χρησιμοποιούμε διάφορες εκφράσεις. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι σε καφενείο. Και μια που έχω το λόγο σχετικά με, την, ε, με το κράτος δικαίου. Η Σλοβακία ανήκει ε, στην ε, ομάδα των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στο άνω μέρος της κλίμακας ε, όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης. Είμαστε μεταξύ των πρώτων 13 χωρών. Και όσον αφορά το κράτος δικαίου, παρετήθηκε ο Πρωθυπουργό μας, έπεσε η κυβέρνηση, υπάρχει μια νέα κυβέρνηση σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα οι ένοχοι συνελήφθησαν και ίσως ε, συμβαίνει αυτό μερικές φορές. Οι εγκέφαλοι να μην συλλαμβάνονται, να μην αποκαλύπτονται. Ε, η Σλοβακία θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Περιμένω να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν άνθρωποι, όπως υπάρχουν και παντού, υπάρχουν και στη Σλοβακία άνθρωποι που είναι διεφθαρμένοι και η διαφθορά δεν είναι πρόβλημα μόνο στη Σλοβακία ή τη Μάλτα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το κατά πόσον η χώρα μπορεί να κάνει κάτι κατά της Σλοβακίας και νομίζω ότι η Σλοβακία το κάνει. Ευχαριστώ. Σοφή, πιέζει ο χρόνος. Έχουμε ξεπεράσει τα γονικά όρια. Αν μπορείς να κλείσεις κατα τη θέμα και μετά να κλεισει το θεμα και μετα να παμε στα συμπεράσματα. Ευχαριστώ Κλώδη και τους συναδέλφους που μίλησαν. Πρώτα πρώτα θέλω να πω ότι κρίμα που έφυγε η κυρία Μπένοβα γιατί με εξέπληξε και με ανησύχησε με τα όσα είπε. Πάντως νομίζω ότι αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια κοινότητα αξιών και κράτους δικαίου, ε, τότε θα πρέπει να προχωρήσουμε. Θα πρέπει να αφήσουμε την ε, αμυντική ενστικτόδη αντίδραση στις επικρίσεις. Δεν επικρίνουμε κάποια χώρα, δεν ε, ε, υποστηρίζουμε το α κόμμα έναντι του β. Θέλουμε το καλό του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όταν κάτι πάει στραβά σε μια χώρα, τότε όλο το σύστημα βλάπτεται. Είδατε τι έγινε και με την εκτέλεση των ε, ενταλμάτων, ε, των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψη. Ε, μα γι' αυτό σας λέω, ας είμαστε λίγο παραπάνω ανοιχτοί στις επικρίσεις συγκεκριμένων θεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αν αφορούν τη δική μας χώρα. Και ήθελα να πω στην δεν πρόκειται περί ψηφίσματος, πρόκειται για μια έκθεση ενδελεχή και τεκμηριωμένη. Είπε η κυρία Μπένοβα ότι αυτές οι εκθέσεις είναι ανακριβείς και με ε, εκπλήσει γιατί ήταν παρούσα. Από πού και που επομένω βρίσκει ανακριβείς τις εκθέσεις. Επίσης, ε, το θέμα δεν είναι δυσκολίες σε συγκεκριμένες σχέσεις ε, κάποιων πολιτικών με κάποιους ε, δημοσιογράφους. Πρόκειται για μια γενικευμένη εχθρική στάση έναντι των δημοσιογράφων. Και τι να σας πω, να λέει κανένα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα όταν κοίται νεκρός ένας δημοσιογράφος. Πρόκειται περί ισχυρισμού απαράδεκτου. Ε, βέβαια υπάρχει πρόβλημα όταν κάποιος ερευνητής δημοσιογράφος που ερευνούσε τη διαφθορά ε, σκοτώθηκε από κάποιον ε, ε, επαγγελματία δολοφόνο που κάποιος ε, ε, τον έστειλε σε αυτή την αποστολή. Ε, αυτή η παρατήρηση είναι πάρα πολύ απρεπής. Ε, βέβαια και νομίζω ότι είναι τεκμηριωμένα όσα λέμε. τώρα για την κυρία Γκόμες και μπράβο της για την προηγούμενη φάση δούλεψε σκληρά. Α, είπατε ε, δύο την το οποία αποδεικνύει ότι είμαστε αμερόληπτοι και ουδέτεροι. Οι ισχυρισμοί του κυρίου Καρντόνα, ε, από ό,τι κατάλαβα, κατέπεσαν. Γιατί απεδειχθήκε ότι αυτός που έκανε αυτούς τους ισχυρισμούς, τα όσα είπε, τα απέσυρε. Να δούμε πόσο θα εξελιχθεί το πράγμα. Φυσικά και θα πρέπει να τα λέμε τεκμηρωμένα, αλλιώ κάνουμε αξιοπιστία. Τώρα για την τηλεόραση. Δεν νομίζω ότι γινόταν έρευνα για την διαφθορά. Απλώ ε, φιλοξένησε για δύο δημοσιογράφου που έκαναν αυτή την έρευνα. Δεν είναι ακριβώ το ίδιο. Αύριο, συνάδελφοι, θα έχουμε αυτή. Θα έχουμε μια κρόση με τρει Βουλγάρους δημοσιογράφου. Οπότε θα έχουμε πληροφορίε από πρώτο χέρι και σα καλώ όλους να έρθετε τώρα. Όσον αφορά την Europol, είχαμε μια σειρά συναντήσεων συναντήσουν από κοντά. Είχαμε και κάποιες τηλεσυνεδριάσεις και μας διαβεβαίωσαν ότι η συνεργασία τώρα πάει πάρα πολύ καλά και τώρα έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται. Εγώ έχω ακόμα κάποια ερωτηματικά, αλλά γενικά ε, χαίρομαι που και στις δύο χώρες ε, οι αρχές είναι πρόθυμες να συνεργαστούν. Φυσικά και ήταν πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της ε, Europol και για το ψήφισμα θέλω να πω ότι θα πρέπει να βαθμιστούν οι αρμοδιότητες της Europol. Θα πρέπει να μην εξαρτάται το τι θα κάνει η Europol από το αν θα προσκληθεί από τις ε, αρχές. Όχι, όχι, όχι κύριε Φράντς, δεν διερευνήσαμε ε, τους ισχυρισμούς, τα όσα διατυπώνονται κατά των ε, ε τσιγκάνων. Για την κυρία Μετσόλα τώρα. Ε, βέβαια και συμφωνούμε ότι χρειάζεται να υπάρχει ένας αντικειμενικός ε, μηχανισμός, η Επιτροπή θα πρέπει να κατεβάσει μια σχετική πρόταση. Επίσης, συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε για το ότι θα πρέπει αυτή η έκθεση να δημοσιοποιηθεί. Την έχει δει ο Πρωθυπουργός. Ε, αφορά την σύζυγό του και αφορά αυτή η έκθεση και μέλη της κυβέρνησης. Άρα θα πρέπει να δημοσιοποιήσει τα γραφόμενα. Ποια είναι ο Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να απαγορεύεται τη δημοσιοποίηση. Δεν, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από το δίκαιο. Είπατε για το κράτος δικαίου, για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Τέλος, κυρία Μακοβέ, είσαστε κάπως ε, απεσιόδοξοι όσον αφορά τις πιθανότητες κάποτε να συλληφθούν ε, αυτοί που βρίσκονται πίσω από τις ε, δολοφονίες αυτές. Όχι, εγώ δεν είμαι τόσο απεσιόδοξη. Και στην Σλοβακία μετά τα αρχικά λάθη της αστυνομίας το ότι συνελήφθησαν οι δολοφόνια είναι θετικό. Θα πρέπει αυτό να το εκτιμήσουμε. Και έχω την εντύπωση ότι συνεχίζονται οι έρευνες και ότι είναι σοβαρές. Συνάντησα πολλούς που είπαν ότι ενδιαφέρονται στα σοβαρά για να υπάρχει ανεξαρτησία, διαφάνεια στην δίκηση. Δεν είναι όλα μαύρα και άραχλα. Και εν πρόεδρε. Α, Κάτι ξέχασα για τον κύριο Νάγκη. ότι θα πρέπει να είμαστε επικριτικοί. πρέπει μάλλον ότι να, να, λάβουμε υπόψη το ότι κάποιοι έχουν ε, Να είμαστε λοιπόν τόσο αυστηροί. Ε, ναι, αλλά από τη μία βγήκανε από κυβέρνηση και αστυνομία, μπορεί να μπουν από την άλλη. Άρα, τέλος πάντων, αποφύγαμε να τα πούμε αυτά όταν ήμασταν στη χώρα. Άρα, συνεχίζουμε την προσεκτική παραγωγή των εξελίξεων. Θα πρέπει να γίνουν επιτόπου επισκέψεις και συναντήσεις, με η Europol και να έρθουμε σε επαφή με όλες τις αρμόδιες αρχές, με ό,τι διαδικασία θεωρείται πιο δόκιμη και όλα αυτά ισχύουν για όλες τις χώρες μέλη της Ένωσης. Αυτά. Λοιπόν, υπάρχει ένα ψήφισμα, μάλλον ετοιμάζει η ομάδα εργασίας ένα ψήφισμα που προβλέπεται για το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τη Σοφία και όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν σε αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα. Λοιπόν, ε, έχουμε καθυστερήσει λίγο, ας προχωρήσουμε. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στο σημείο 10. Πρόκειται ε, για τον κανονισμό που αφορά την αποτελεσματική και αποδοτική συνεργασία μεταξύ της Όλαφ και όλων των άλλων οργανισμών για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της κοινότητας. Η Μόνικα Μάκαβη είναι η συγγήτρια, έχει το... Ε, ε βρίσκεται εδώ η κυρία Μάκαβη, θα της δώσω το λόγο αμέσως. If, you, if you're leaving uh, now, please Thank you. Η κυρία Μάκαβη, παρακαλώ. Ευχαριστώ σχεδόν 20 χρόνια μετά την ε, ίδρυση της Όλαφ, κάνουμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Το βήμα αυτό είναι η δημιουργία του, της Ευρωπαϊκής εισαγγελία. Είναι πολύ σημαντικό τώρα να, τον, να, να θεσπιστεί και να ενισχυθεί ο μηχανισμός και να δοθούν σαφείς κανόνες για το μηχανισμό της συνεργασίας ανάμεσα στην Όλαφ και το EPPO, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλοί σαφείς κανόνες για το ποιος κάνει τι. Αυτή η στενή συνεργασία πρέπει να βασίζεται στις αρχές της συμπληρωματικότητας, της μη επικάλυψης και της ανταλλαγής πληροφοριών η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διεξάγει τις ε, ε, ποινικέ έρευνες ε, και διώξεις, ενώ η Όλαφ θα έχει την ευθύνη μόνο για τις διοικητικές έρευνες που σχετίζονται με τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό η σχέση ανάμεσα στην Όλαφ και την Εισαγγελία, την Ευρωπαϊκή, να μην δημιουργεί διαμάχες όσον αφορά τον καταμερισμό των ε, αρμοδιοτήτων. Ε, θα πρέπει ε, να μην ε, διεξάγουν και οι δύο οργανισμοί έρευνες για τα ίδια γεγονότα. Χρειάζεται υψηλή προστασία ε, των δεδομένων και εμπιστευτικότητα και γι' αυτό πιστεύουμε ότι όλα θα πρέπει να έχει έμεση πρόσβαση ε, στο σύστημα μέσω ενός ατόμου που θα έχει οριστεί από την ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα για τη μη επικάλυψη των ερευνών, η όλα θα πρέπει να ενημερώνει αμέσω την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για οποιοδήποτε εγκληματική δραστηριότητα όπου θα έχει αρμοδιότητα η εισαγγελία και δεν θα πρέπει να ανοίγει έρευνε για θέματα που ήδη ερευνώνται από την ΕΠΠΟ. Βέβαια, αν δώσει διαφορετική εντολή η ΕΠΠΟ, η Όλαφ θα πρέπει να ακολουθεί αυτές τις εντολές, αυτές τις οδηγίες. Αν η εισαγγελία ε, οι περισσότερες πληροφορίες για ε, κλιματική συμπεριφορά που εντοπίζει η Όλαφ, ε, θα πρέπει να ε, υπάρχει σχετική συνεργασία. Στην περίπτωση που η εισαγγελία ήδη διεξάγει ποινική έρευνα και ε, ο Γενικός Διευθυντής της Εισαγγελίας θεωρεί θα πρέπει να ανοίξει ε, η έρευνα και να ε, διεξαχθεί ίσως από την Όλαφ, αυτό θα πρέπει να γίνεται με επίσημη άγκριση από την Εισαγγελία. Στην περίπτωση ποινικών ερευνών δεν θέλουμε αυτές να τίθενται σε κίνδυνο λόγω των διοικητικών ερευνών που γίνονται παράλληλα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ε, ε, τα ευρήματα των ερευνών να γίνονται ε, αποδεκτά από το δικαστήριο. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, τηρούνται όλες οι απαραίτητες ε, διασφαλίσεις και εχέγγυα. Η Όλαβ δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το πεδίο των διοικητικών ερευνών, γιατί στην περίπτωση αυτή είναι σαφές ότι τα ευρήματα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα δικαστήρια. Και δεν θέλουμε να γίνεται κάτι τέτοιο. αν η εισαγγελία μπορεί, θέλει να ζητήσει η Όλαφ να συμπληρώσει το έργο της στην περίπτωση ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, ιδίως στα πλαίσια του άρθρου 12ε, ε, μπορεί η εισαγγελία να αναθέσει ε, το έργο αυτό στην Όλαφ, χωρίς να διακυβεύεται η δική της ε, δράση. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία μπορείτε να βρείτε στην γνωμοδότησή μου. Ίσως θα πρέπει να πω ότι για τα κράτη-μέλη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το ερώτημα είναι τι θα γίνει με αυτά τα κράτη-μέλη. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η απάντηση είναι ότι η Όλαφ θα συνεχίζει να κάνει ό,τι έκανε μέχρι τώρα και όταν ε, υπάρχουν ε, ε, ποινικές έρευνες ή έρευνες για, για, για εγκληματικές δραστηριότητες θα πρέπει να αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές. Και όταν υπάρχουν ποινικά δικήματα οι άνθρωποι θα παραπέμπονται στην χώρα καταγωγής τους. Νομίζουμε ότι στην περίπτωση αυτή δεν, υπάρχουν άλλοι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να χειριστούμε αυτές τις υποθέσεις. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι μέχρι τις 26 Νοεμβρίου. Λοιπόν, είναι σχέδιο γνωμοδότηση αυτό που συζητάμε. Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου υπάρχει προθεσμία για υποβολή τροπολογιών, λέει ο Πρόεδρος. Ε, θα ήθελε κανείς να πάρει το λόγο για το θέμα αυτό ή να κάνει ερωτήσεις. Όχι. Αν όχι, ευχαριστώ την ε, κυρία συνάδελφο για την ε, Μάκαβη. Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου είναι, όπως είπαμε, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα 21 της ημερήσης διάταξης. Okay, so have, um, the... είναι ο κύριος Ράντεφ. Έχουμε κάποιες τροπολογίες για την έκθεση αυτή σχετικά με τους κανόνες που διευκολύνουν τη χρήση χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, εντοπισμό, έρευνα και δίωξη κάποιων εγκληματικών πράξεων. Ε, ο κύριος Ράντεφ νομίζω ότι θα πάρει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ομιλώ εξ ονόματος ε, του κύριου Ράντεφ, ο οποίος ψηφίζει στην Επιτροπή ε, Νομικών Θεμάτων και ε, δυστυχώς κολλείεται. Ο εισηγητής χαίρεται για τις 150 τροπολογίες που έχουν καταθέσει και οι οδησηγητές. Αύριο θα συναντηθούν οι σκιώδεις εισηγητές με τον εισηγητή. Οι περισσότερες από τις τροπολογίες βρίσκονται μέσα στο συνολικότερο πλαίσιο της έκθεσης. Είναι σημαντικό για τον κύριο Ράντεφ να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών. Η ψηφοφορία σχεδιάζεται για την 3η Δεκεμβρίου. Ο δε κύριος Ράντεφ είναι πεπισμένος ότι η έκθεση θα εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία. Μάλιστα, στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου όπου θα συζητηθεί. Uh, Σα ευχαριστώ πολύ κύριε ε, συνάδελφε ε, που λάβατε το λόγο εκ μέρους του κύριου Ράντεφ. Η κυρία Τσινίτσι θέλει να ε, τοποθετηθεί αλλά είναι εδώ. θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα και μάλιστα ταχαίως, αν δεν θέλει κανείς άλλος. Υποθέτω ότι κανείς άλλος δεν θέλει να παρέμβει. E Ποια είναι η προβλεπόμενη ώρα αφήξης της κυρίας Τσινίτσι, το πω έτσι. χρειαστεί λοιπόν να προχωρήσουμε τότε, γιατί είναι άγνωστο πότε ακριβώ θα προσέλθει. Εκτό αν κανεί άλλο θέλει να ομιλήσει. Α, η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή. Καλώ. Θέλετε να πείτε δύο λόγια εσείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Λίγα λόγια. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι απόντες οι περισσότεροι σκιώδεις συγητές, αλλά μπορώ να πω κάτι που θεωρώ σημαντικό. Σας ευχαριστώ που ε, προσφέρατε, που δεχτήκατε μάλλον κατεπηγόντα χαρακτήρα για τη συζήτηση αυτή. Αρχίζουμε τους τριμερείς διαλόγους στον Δεκέμβριο, αν αυτό είναι δυνατόν, και να ολοκληρωθεί η έγκριση μέχρι τον Απρίλιο, όσο θα υπάρχουν ολομέλειες ακόμη δηλαδή. Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα, το οποίο μας ανησυχεί, για το άρθρο 7 της προτάσεως, το οποίο αναφέρεται σε καταστάσεις όπου όργανα επιβολής του νόμου ζητούν πληροφορίες από Financial Intelligence Units και αυτά περιλαμβάνονται στην τέταρτη οδηγία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που λέει ότι η FIU θα πρέπει να μπορεί να τα αποκρίνεται σε αιτήσει των αρχών επιβολή του νόμου για χωρί κυκλοφοριών. Στην πρότασή μα προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία αυτή, απαιτώντα από την FIU να συμμορφωθεί με τα αιτήματα αυτά των αρχών επιβολή του νόμου. Βλέπουμε ότι το Κοινοβούλιο έχει καταθέσει, οι περισσότερε δηλαδή πολιτικέ ομάδε έχουν καταθέσει τροπολογίε απόρριψη τη ιδέα αυτή για να επανέλθουν στο is entitled to reply. Τονίζω ότι αυτό σημαίνει δεν θα υπάρξει ενίσχυση της ε, εφαρμογή των, των διατάξεων. Και αυτό μας ανισχύει πολύ, διότι ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους καταθέσαμε την πρόταση είναι λόγω των επανειλημμένων ετοιμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την, και μιλώ για την έκθεση της Πάναμε Κομίτη του κ. Νάρτ από τον Φεβρουάριο, όπου ζητήσατε ξανά και ξανά ενίσχυση της ισχύω των κανόνων. Δυστυχώς η διατύπωση των τροπολογιών δεν ενισχύουν τους κανόνες αυτούς. Τους κρατούν στο ίδιο επίπεδο. Εμείς θεωρούμε ότι οι κανόνες πρέπει να είναι πλέον ισχυροί και γι' αυτό σας παρακαλούμε να επανεξετάσετε την θέση που λαμβάνετε μέσω των τροπολογιών σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Θα μεταφέρουμε το σημαντικό αυτό μήνυμα στα αρμόδια πρόσωπα. Ε, ευχαριστώ και ευχαριστούμε εμέσω και τον κύριο Ράντεβ. Ο κύριος Λετζέρι του Frontex έχει καθυστερήσει λίγο. μα μένει λίγος χρόνος μέχρι να, ε, μέχρι να καταφτάσει για το επόμενο θέμα. Άννα Γκόμε, ζητήσατε το λόγο αν θέλετε να τοποθετηθείτε διαβραχιών. Ναι, σχολιάζω τα όσα ακούσαμε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρωτοβουλία και για την προειδοποίηση που μας απευθύνει για την λυπηρή αυτή εξέλιξη που έχουν προκαλέσει ορισμένα μέλη. Ένα είδος οργάνωση με ύποπτους ε, σκοπούς φαίνεται να κρύβεται από πίσω για να ανατρέψει ένα αίτημα το οποίο είναι διαρκές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και χρηματοδότηση τρομοκρατίας με την Ευρωπαϊκή FIU. Ευχαριστώ ιδιαίτερα λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αξίζει την πλήρη υποστήριξη των Ευρωβουλευτών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σε ό,τι αφορά τη δική μου πολιτική ομάδα, επανεξετάζουμε αμέσως τα όσα έχουν συζητηθεί για να είμαστε βέβαιες και βέβαιοι ότι παραμένουμε εντός των πλαισίων της βασικής αυτής αρχής μάλλον τη βασική αυτή γραμμή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τον συνάδελφό μα που ε, έλαβε το λόγο εκ μέρου του κ. Ράντεφ και που θα μεταφέρει τα μηνύματα αυτά στον ίδιο τον κ. Ράντεφ. Θα εγκριθεί το σχέδιο χθε μέχρι τι 3 Δεκεμβρίου. Και ε, προχωρούμε στο επόμενο μέχρι ε, ότου καταφτάσει ο κ. Λετζέρη, που μπορεί να πάρει λίγα λεπτά ακόμη για να συζητηθεί το επόμενο θέμα, δηλαδή 22 Frontex. Ξαναλέω, αναμένουμε τον κύριο Φαμπρίς Λετζέρη. Ε, τότε ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα λίγων λεπτών. Uh, um, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Έχουμε τον κύριο Λετζέρη κοντά μας. Προχωρούμε στο υπαριθμό 22 της ημερησίας διατάξεως, που είναι το θέμα που αναφέρεται στον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Η Επιτροπή μας συντάσσει την ε, γνωμοδότησή της για τη, μάλλον τη θέση της για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για να μας βοηθήσει στην προπαρασκευή αυτή απευθύνω το καλό ορίσατε τον κύριο Λετζέρη που είναι εκτελεστικός διευθυντής του Frontex και θα αναπτύξει τα σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2017 σε εφαρμογή του κανονισμού 656-2014 για την προστασία των συνόρων. και βεβαίως μπορείτε να τον ερωτήσετε ό,τι θέλετε για θέματα που σας ενδιαφέρουν ε, από αυτό το δραστηριοτήτων του σημαντικού αυτού οργανισμού. Κύριε Λτζέρη, λοιπόν, σας παρακαλώ, ε, ε, μπορείτε να λάβετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές. Ο σκοπός της παρέμβασής μου είναι να σας αναφέρω τις τρέχουσες δραστηριότητες του Frontex. Η έκθεση για το 2017 έχει δημοσιευτεί, αλλά θα ήθελα να σας ενημερώσω και για τις τρέχουσες δραστηριότητες. Γενικά νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι τώρα έχουμε μια ενισχυμένη ε, εντολή. Μιλάω για αυτή που δόθηκε το 2016, όχι για μελλοντικές προτάσεις, μιλάω για την τρέχουσα εντολή. Ε, έχουμε, από ό,τι φαίνεται, ε, περισσότερες δυνατότητες, σύμφωνα με την εντολή αυτή, αλλά και περισσότερους πόρους στη διάθεσή μας. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και είναι σημαντικό είναι ότι ίσως στο παρελθόν ο οργανισμός μας γινόταν αντιληπτός κυρίως ως ένας φορέας που, το, που ασχολόταν μόνο με θέματα μετανάστευσης. Αλλά πρέπει να πω ότι η διαχείριση των συνόρων δεν αφορά μόνο τη μετανάστευση. Υπάρχουν όλο και περισσότερα θέματα που αφορούν την ε, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ή την πρόληψη της τρομοκρατίας και μερικές φορές αυτά τα θέματα ε, αποσυνδέονται από τα θέματα της μετανάστευσης και νομίζω δεν δε σχετίζονται. Και επίσης είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι το πεδίο δράσης του Frontex θα πρέπει να είναι όσο ευρύ είναι το θέμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων. Να σας δώσω ορισμένα στοιχεία. Τους πρώτους δέκα μήνες της φετινής χρονιάς ο αριθμός των παράνομων διαλεύσεων, διαλεύσεων ε, μειώθηκε κατά 30% των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύγκριση με την κατάσταση που αντιμετωπίζαμε πριν από ένα χρόνο. Συνολικά καταγράψαμε φέτος περίπου 120.000 παράτιμες διαλέψεις των συνόρων. Η κατάσταση αυτή οφείλεται κυρίως στις μικρότερες μεταναστευτικές πιέσει στη Νότια Μεσόγειο και οι μεγαλύτερε αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Δυτική Μεσόγειο και στα χερσαία σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα, αλλά τα απόλυτα νούμερα εδώ ε, παραμένουν σχετικά χαμηλά. Αυτό σημαίνει ότι προ το παρόν από επιχειρησιακή σκοπιά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή η μεταναστευτική κρίση στα εξωτερικά σύνορα. Παρακολουθούμε την κατάσταση, υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη, αλλά η στιγμή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να σκεφτούμε στρατηγικά πώς μπορούμε να ε, εξελιχτούμε στο μέλλον. Ανέφερα το γεγονός ότι η διαχείριση των συνόρων δεν αφορά μόνο τα θέματα της μετανάστευσης. Ήθελα να πω ότι πρόσφατα ε, υπήρξε μια κοινή δήλωση αλλά και μια κοινή αξιολόγηση ε, Europol και Frontex σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων σχετικά με την ενίσχυση της ενεργασίας μας. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η ακτοφυλακή γενικά η συνοριοφυλακή γενικώ, αλλά και ο Frontex ε, ε, ε έχουν κοινέ επιχειρήσεις σε επίπεδο συνόρων και μπορούμε να είμαστε τα μάτια και τα αυτιά ε, των ε, αρχών επιβολής του νόμου, ούτως ώστε να μπορούμε να τροφοδοτούμε τις αρχές των κρατών μελών με τα δεδομένα που συλλέγουμε από τις δραστηριότητές μας. Εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι για έρευνες, αλλά ε, οι συνοριοφυλακές και στα κράτη-μέλη ε, μπορούν ε, να συλλέγουν ε, στοιχεία για εγκληματικές δραστηριότητες που τροφοδοτούν τις έρευνες για τις εγκληματικές αυτές δραστηριότητες. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι είμαστε όλο και περισσότερο ε, επιχειρησιακοί, ε, ε, έχουμε περισσότερες επιχειρησιακές δυνατότητες, λειτουργούμε 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να επιχειρούμε η μέρα και νύχτα ανα πάσα στιγμή και μπορούμε να ενισχύουμε και τη δράση των κρατών μελών στα εξωτερικά σύνορα. Έχουμε και κάποιες παραδοσιακές κοινέ επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ο μέσος όρος του μεγέθους των επιχειρήσεών μας είναι περίπου 1.500 αξιωματικοί ε, και ενώ και συνοριοφύλακες βέβαια αλλά και ακτοφυλακοί σε σκάφη 1.500 άτομα, 1.500 αξιωματικοί φαίνεται να είναι, το, να είναι ο μέσος όρος όταν δεν υπάρχει ενεργοποίηση του συστήματος Rapid Intervention. Έχουμε τρεις μεγάλες επιχειρήσεις. Ποσειδών στην Ελλάδα, ε, Θέμης στην Ιταλία, η οποία επιχείρηση τροποποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2018 με ένα στοιχείο περισσότερο ασφάλειας και επιβολής του νόμου για να λάβουμε υπόψη μας και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών που παρατηρήθηκε μεταξύ Αλβανίας και Ιταλίας καθώς επίσης και το λαθρεμπόριο όπλων μερικές φορές. Και έχουμε, και αυτό είναι η καινοτομία της ε, ε, χρονιάς αυτής, ε, ότι έχουμε ε, μια επιχείρηση στα νότια της Ισπανίας, γιατί η ροή από το Μαρόκο προς την ε, Ισπανία τεταπλασιάστηκε και πενταπλασιάστηκε τα τελευταία τρία χρόνια. Θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την έρευνα και διάσωση, και αυτό είναι μέρος των θαλάσσιων επιχειρήσεων. Μέχρι τώρα, το 2018, έχουμε σώσει 30.000 ανθρώπους σε όλα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμβάλαμε στην καταχώρηση, στη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και στο screening των ε, νέων αφήξεων. Επίσης συμβάλαμε στη σύλληψη λαθρο, ε, λαθρεμπόρων, συγγνώμη, ε, διακινητών ανθρώπων, καθώς επίσης και κάθε μορφής άλλη παράνομη δραστηριότητα. Πέρυσι, να σας πω ότι συμβάλαμε στη σύλληψη 744 διακινητών ανθρώπων και πάνω από 2.000 ε, ε, ε, λαθρεμπόρων και στην ανακάλυψη 136.000 τόνων ναρκωτικών. Επίσης, θα ήθελα περισσότερο να εστιάσω τώρα στις θαλάσσιες δραστηριότητες και στην θαλάσσια συγκοινωνία. Θα θυμάστε ίσως ότι η νέα εντολή προέβλεπε τριμερή συνεργασία μεταξύ του Frontex, της ΕΜΣΑ και της ΕΦΚΑ. Ε, αντίστοιχα, ε, του Μέσου για τη Θάλασσα και το Ταμείο Αλίας και Θάλασσας. Με αντίστοιχες εντολές ε, λειτουργούν οι τρεις οργανισμοί. Και αυτό εφαρμόζουμε τώρα με πολύ θετικά αποτελέσματα στις επιχειρήσεις μας και στις δραστηριότητές μας. Όσον αφορά την έρευνα και ε, διάσωση αλλά και την καταπολέμηση της παράνομης αλίας αλλά και επίσης τη συνεισφορά μας στην καταπολέμηση ε, της ε, ρήπανσης αλλά ακόμα και του περιβαλλοντικού εγκλήματος. Η βασική ιδέα εδώ είναι ότι οποτεδήποτε υπάρχει ένα σκάφος που κάνει περιπολίες, είτε είναι της Frontex είτε του ΕΦΚΑ, το πλήρωμα Μερικές φορές μάλιστα έχουμε και ε, επιθεωρητές αλίας στα σκάφη μας, ε, γιατί πρόκειται για περιπολίες πολλαπλών σκοπών. Ε, αυτοί λοιπόν που βρίσκονται πάνω στο σκάφος, όποια και είναι η ιδιότητά τους, μπορούν να υποβάλουν αναφορά στον Frontex, είτε για σκάφος που μεταφέρει παράτυπους μετανάστες ή να αναφέρει περίπτωση ρήπανσης ή παράνομης αλίας. Κατά τη γνώμη μου, από αυτά που μαθαίνουμε, αυτό το μοντέλο τριμερού συνεργασίας μεταξύ των τριών θαλάσσιων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εξελίσσεται σε πραγματικά βέλτιστη πρακτική και ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, και σε άλλους τομείς δραστηριοτήτων. Ο τρόπος αυτός λειτουργίας εξασφαλίζει ότι ε, η ακτοφυλακή ε, των κρατών μελών ε, αισθάνεται ότι μπορεί να ενσωματωθεί σε αυτές τις δραστηριότητες και πρέπει να σας πω ότι έχει διαπιστωθεί ότι έχουν ευθυγραμμιστεί οι προτεραιότητες του Φόρουμ των Ευρωπαίων Αυτοφυλακών και ε, ε, με, με, το στόχο αυτών των τριών ευρωπαϊκών οργανισμών. Αυτό με φέρνει στον κανονισμό 656 56 του 2014 ε, ε, ε, εκδόθηκε μια ειδική έκθεση προς το Κοινοβούλιο φέτος τον Ιούλιο. Αυτός είναι ο κανονισμός που θεσπίζει τους κανόνες για την εποπτεία των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στα πλαίσια των επιχειρήσεων του Frontex. Οι κοινέ επιχειρήσεις που είναι αντικείμενο ε, αξιολόγηση στα πλαίσια αυτής της έκθεσης είναι ο τρίτον πριν από το Θέμη στην Ιταλία, Ποσειδών στην Ελλάδα, ε, Ιντάλο στην Ισπανία, συν άλλη μια ε, που επίσης φιλοξενεί η Ισπανία ε, μεταξύ ε, των Καναρίων και της ε, Αφρικανικής ε, ακτής. Ο, σκοπός του Frontex είναι πάντοτε να υπάρχει προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με τα δικαιώματα αυτά και υπάρχει ο αξιωματικός που είναι υπεύθυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και που η γνώμη του επισυνάπτεται σε αυτή την έκθεση. Τώρα, για την αποβίβαση σε τρίτες χώρες. Στη φάση της προετοιμασίας του επιχειρησιακού ε, σχεδίου υπήρχε τέτοια πρόβλεψη για το Ποσειδόνιο, για το Ήρα, παραδείγματο χάρη, την επιχείρηση Ήρα, το 2017. Κατά την ε, φάση της προετοιμασίας του επιχειρησιακού σχεδίου, το, ο Frontex ζήτησε από το φιλοξενούν κράτος μέλος να δώσει μια γενική αξιολόγηση ε, της κάστοτε τρίτης χώρας για την οποία πρόκειτο. Παρόλο που αυτό ήταν ένα θέμα συζήτησης μεταξύ του Frontex και της Ευρωπαϊκής Ένωση και κάποιων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωση που φιλοξενούσαν τις επιχειρήσεις, οι αποβιβάσει σε τρίτες χώρες δεν έλαβαν χώρα στα πλαίσια των κοινών αυτών επιχειρήσεων του Frontex και υπάρχει μια κατάσταση που νομίζω ότι είναι σημαντική και είναι η εξής. Παράλληλα με αυτές τις ε, κοινέ επιχειρήσεις, ο Frontex ανέπτυξε μια νέα υπηρεσία που είναι ε, αέρια υποπτία πολλαπλών στόχων. Αυτό σημαίνει ένα αεροσκάφος που μπορούμε να νοικιάσουμε και με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εποπτεία των συνοριακών ε, δραστηριοτήτων. Αλλά στην περίπτωση αυτή ποτέ δεν μοιραζόμαστε τις πληροφορίες με τις τρίτες χώρες, παρά μόνο με, την, ε, το κράτος μέλος που φιλοξενεί την επιχείρηση ή τις γειτονικές προς αυτό χώρες. Αυτά στα πλαίσια του κανονισμού 656 του 2014. Παρόλα αυτά, και αυτό είναι ένα ερώτημα ίσως για το μέλλον, ε, και λαμβάνοντα υπόψη το γεγονός ότι στην πρότασή τη η Κομισιόν πρότεινε να διευρυνθεί το ε, πεδίο του Eurosur, ε, κάποια στιγμή λοιπόν, ίσως ο Ευρωπαίος νομοθέτης θα πρέπει να σκεφτεί έναν μηχανισμό ο οποίος θα έδινε είτε το πράσινο φως είτε θα απαγόρευε την μετάδοση σε πραγματικό χρόνο των ε, ε, πληροφοριών στις γειτονικές τρίτες χώρες. Θα μπορούσε αυτό να αφορά ε, διάφορες περιπτώσεις ερευνών ή ε, επιβολής του νόμου. Και άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε ε, να ανταλλάξουμε πληροφορίες με τρίτες χώρες σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, η αξιολόγησή μας ως υπηρεσίας κατέληξε στο ότι οι χώρες μέλη ως προς τις γειτονιάς στις τρίτες χώρες ε, ότι θα μπορούσαμε εκεί να έχουμε καλύτερη ρύθμιση του, του, του, του δικού μας καθήκοντος γιατί υπάρχουν πολλές ελλείψεις και τελικά καταλήξανε στο ότι υπάρχει πρόβλημα στην επαφή με τις τρίτες χώρες όσον αφορά τις επιχειρήσεις μας. Για να δούμε τώρα κάτι άλλο. Την συνεργασία στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς. Η αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών σύνορων δεν μπορεί να ξεκινά από τα σύνορα καθε αυτά, αλλά είναι κάτι ευρύτερο. Έχουν να κάνουν δηλαδή και χώρες προέλευσης, χώρες ε, διέλευσης, ίσως και υπάρχουν και κάποιες ε, περιπτώσεις που δεν είναι θέμα μετανάστευση αλλά είναι θέμα καταπολέμησης του διεθνούς διασυνοριακού εγκλήματο. Έχουμε εντατικοποίησει τη συνεργασία μας, όπως λέμε στο κείμενο. Έχουμε και το Africa Frontex Intelligence Community για να έχουμε κάποια τέτοια σχέδια ε, τα οποία έχουν από την ε, Γενική Διεύθυνση της ΔΕΦΚΟ όσον αφορά το σχέδιο της τεχνικής αρχής Και έτσι μπορούμε να επεκτείνουμε τη δράση μας με τη συνεργασία αυτή στις ε, αφρικανικές χώρες και όχι μόνο. Επίσης έχουμε αναπτύξει ε, αυτό το δίκτυο των αξιωματικών συνδέσμων Δυτικά Βαλκάνια, με έδρα το Βελιγράδι, στον Ιεμέη, άλλος για να καλύψει τον Νίγηρα. Τώρα θέλουμε να διευρυνθεί αυτό το δίκτυο στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και στην Αφρική. Όσον αφορά τώρα αυτούς τους αξιωματικούς παλίλους συνδέσμους και τη δουλειά τους εκτός ε, του αρχηγείου. Τώρα αυτοί έχουν αναπτυχθεί στις χώρες συνδεδεμένες με το Σέγγεν, στις χώρες μέλη, σύμφωνα με τον κανονισμό του 16 και έχουμε μέχρι τώρα εκπαιδεύσει 11 τέτοιους ε, υπαλλήλου ε, αξιωματικού Αυτοί έχουν αναπτυχθεί και οι υπόλοιποι όσοι δεν έχουν πάει θα αναπτυχθούν του χρόνου άλλο θέμα τώρα, επιστροφές, επαναπατρισμός, άλλο θέμα το οποίο μας επισχόλησε το 17 αλλά και το 18 ως υπηρεσία. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, λέει ο πρόεδρο τον κύριο Λετζέρη, μέχρι τις 12. Καλά, να σας τα πω πιο συνοπτικά, γιατί προς το παρόν έχουμε τις προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις, αλλά να βλώνουμε και δικά μας αεροπλάνα για, τις, ε, για τον επαναπατρισμό. Πέρσι έκαναμε 341 πτήσεις για τους 14.000 παράνομους μετανάστες που επαναπατρίσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτες χώρες, δηλαδή το 10% των επαναπατρισμών από Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτες χώρες. Κάτι άλλο για τα δημιουργικά διαπιστώθηκε ότι η δράση του οργανισμού σε αυτό τον τομέα έχει θετικές επιπτώσεις όσον αφορά πολλές πτήσεις οι οποίες εποπτεύονται από τους αρμοδίους. Θετική επιπτώση αυτή γιατί ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν υπάρχει τέτοιο αντίστοιχο σύστημα. Τώρα πάλι όσον αφορά την αξιολόγηση της κινητικότητας και αυτό ήταν η νέα μας αρμοδιότητα έχουμε τώρα για δεύτερη χρονιά σερή ε, αυτή την αξιολόγηση της κινητικότητας. Αφορά το πόσο έτοιμα είναι προς τούτο τα κράτη-μέλη αλλά και τον προγραμματισμό. Οπότε τώρα τα κράτη-μέλη ξέρουν τις δυνατότητές τους αλλά επίσης διαπιστώνουμε ότι χρειάζεται το πώς θα υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες. Συγκεκριμένα. Επισημάνθηκε ότι σε καποια κρατημέλη που είναι στα σύνορα της Ένωσης έχουμε κατάσταση ενισχυτική όσον αφορά την φιλοξενία των παρνόμων μεταναστών. Α, και τελικά υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τους ελέγχους στα σύνορα. Από τότε που άλλαξε η Σέγγεν ούτως ώστε να έχουμε υποχρεωτικούς ελέγχους για όλους τους επιβάτες. Επομένως, πρέπει, πρέπει να κλείσουμε στις 12 ε, δεν ξέρω είναι δυνατόν γιατί πολλοί θα έχουν να συμβάλλουν στη συζήτηση οπότε παρακαλώ να βάλουμε τελεία σε αυτό το σημείο να ακούσουμε αυτές τις ερωτήσεις και να σας ε, ξαναακούσουμε. Ε, και εσείς πάλι θα μπορούσατε να ε, συμπληρώσετε όσο έχετε να πείτε και γράφω τώρα για τη Λιβύη. Τι έγινε με το, με το πλοίο τώρα που έχει αυτούς τους 70 επιβάτες που δεν θέλουν να γυρίσει πίσω λόγω της κατάστασης εκεί. Όλα αυτά που μαθαίνουμε για τη Λιβύη Εσείς τι πιστεύετε. Πώς αξιολογείτε τη διαχείριση που κάνουν οι Λίβοι. Τι γίνεται με το DCIM. Έχουμε πληροφορίες. Οπότε αν μπορείτε σχολιάστε και αυτό. Για να δούμε τώρα. Ο κύριος Κόλλιο που είναι ο εισηγητής. Και μετά οι άλλοι που ζήτησαν το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Λετζέρη που ήρθε σήμερα στην Πίμπε. Η ε, επιτήρηση των συνόρων είναι πολύ μεγάλη σημασία διότι επιτρέπει και στο Κοινοβούλιο να αντιληφθεί για ποιο λόγο πεθαίνουν οι άνθρωποι στη Μεσόγειο. Και πολύ σημαντικό διότι οι οδοί προς την Ιταλία γίνονται, η οδός μάλλον προς την Ιταλία, εδώ εισαγωγικών η οδός γίνεται όλο και πιο θανατηφόρα. Και αυτοί οι τελευταίοι μήνε είχαν τα περισσότερα θύματα, το οποίο με οδηγεί στην πρώτη μου ερώτηση για την επιχείρηση τρίτων. Η έκθεσή σας λέει ότι οι περισσότερες διασώσεις έγιναν με τα asset από την επιχείρηση Σοφία και από μη κρατικέ οργανώσεις. Γιατί? Μπορείτε να δώσετε ακριβείς αριθμούς ή ποσοστά, 80%, 70%. Πόσα ήταν με ευθύνη των NGO και πόσα ήταν με την ευθύνη της επιχείρησης Σοφία. Δεύτερο, τα μέτρα που έλαβε η σημερινή Ιταλική κυβέρνηση κατά τον NGO, τι επιπτώσει είχαν. Κάτι άλλο. Ω εισηγητή για τον κανονισμό, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο με το κείμενο που ισχύει. Ήμουν και πριν από τέσσερα χρόνια και τώρα πάλι είμαι ικανοποιημένο. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεσή σα, ο οργανισμό σα που έχει λάβει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση από ποτέ, θεωρεί ότι υστερεί απέναντι σε εθνικέ αρχέ και σε ορισμένου άλλου οργανισμού. Είμαι βέβαιος ότι αυτό που θεωρείτε και εσείς είναι ότι πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και να μην μειωθούν τα πρότυπα, τα στάνταρντ. παρόλο που ενδέχεται να αποτρέπει τις ε, αρχές από του να επιτρέπουν αποβίβαση σε τρίτες χώρες. Και τέλος, είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσουμε ότι το τρέχον ιστορικό είναι διαφορετικό από τότε που εγκρίθηκε ο κανονισμός. Το τωρινό δηλαδή ε, περίγραμμα ας πούμε το background. Όμως η αλλαγή του background δεν δικαιολογεί μείωση των υποχρεώσεων Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης όπου αυτές είναι αναγκαίες. Ευχαριστώ πολύ Κάρλος πολύ σύντομη παρακαλώ. Παρακαλώ δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο, αλλά παρακαλώ να, ε, να παραμείνετε μέσα στα δύο λεπτά. Ορίστε. Ναι, εσείς. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, αλλά αρχίσαμε με καθυστέρηση. Και αυτό βεβαίως είναι ενοχλητικό για όλους, το καταλαβαίνω. Ορίστε λοιπόν, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, φίλε Πρόεδρε. Κύριε Λετζέρη, ευχαριστώ για την έκθεσή σας. Είναι γνωστές οι καταστροφικές συνθήκες στους καταβλισμούς της Λιβύης και καταστροφικές συνθήκες που επιβεβαιώνονται από πολλές παρτυρίες με θανάτους, με βιασμούς Δεν υπάρχουν επανεισδοχές πλέον ε, προσφύγων από σκάφη του Frontex. Τώρα οι πλατφόρμες αποβίβασης συζητούνται τώρα και η ερώτησή μου είναι ο Frontex είναι διατεθειμένος στην εφαρμογή της ιδέας αυτής των πλατφορμών αποβίβασης να τους επαναφέρει στη Λιβύη και δεύτερο θεωρεί ο Frontex ότι πρόσφυγες οι οποίοι έχουν κολλήσει στη Λιβύη θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε προστασία ή και σε καθώς ασύλου και πώς πρόσωπα εξάλλου τα οποία βρίσκονται σε καταλόγους κυρώσεων του ΟΗΕ εξακολουθούν ε, να επανδρώνουν επισήμως ε, τις ακτοφυλακές όπως για παράδειγμα ο Μοχάμετ Κάχλαφ και με ποια κριτήρια ο Frontex επιλέγει με ποιον συνεργάζεται για παράδειγμα σε εκπαιδεύσεις και έχει υπάρξει κάποιο στοιχείο διαφάνειας εν προκειμένου. Άλλη ερώτηση για τρίτες χώρες όπως η Τινησία Θεωρεί ο Frontex ότι η Τινησία μπορεί να θεωρηθεί place of safety σύμφωνα με το Διεθνές Θαλάσσιο Δίκαιο. Θεωρεί ο Frontex ότι σε περίπτωση επανεισδοχής στην Τινησία διατηρείται το δικαίωμα για έξοδο από την χώρα και σύμφωνα και με τη συνθήκη της Γενέβης ε, γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των προσφύγων και τέλος για την εντολή ε, του Frontex στη Μεσόγειο. Ναι, ολοκληρώστε, λέει ο πρόεδρος. Στα πλαίσια της διεύνησης των αρμοδιοτήτων του θεωρεί ο Frontex ότι μπορεί με τα σκάφη του όχι μόνο να φυλάσει τα σύνορα, αλλά να διασώζει ανθρώπινες ζωές περισσότερο με τα σκάφη αυτά. Okay, thank you. Colleagues, a maximum... Ευχαριστώ. Το πολύ δύο λεπτά, αλλιώς δεν θα υπάρχει χρόνος για απαντήσεις. Έλλη Σλάιν. Για δύο λεπτά, το πολύ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Διευθυντή. Ήθελα να κάνω τρεις ερωτήσεις πολύ γρήγορες στον ε, κύριο Λετζέρη. Πρώτον, πόσες επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποίησε ο Τρίτον το 2018, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία του UNCHR έγινε πιο επικίνδυνη η αδρομή στην κεντρική Μεσόγειο και ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε ε, τους μήνες αυτούς και για κάθε 18 άτομα υπάρχει ένας νεκρός, σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές. Πόσες επιχειρήσεις διάσωση πραγματοποίησε ο τρίτον ε, φέτος. Δεύτερη ερώτηση. Είστε παρόντες ως Frontex στα σύνορα μεταξύ Βοσνίας, Ερζεγοβίνη και Κροατίας, γιατί οι οργανώσεις που λειτουργούν επί τόπου μα καταγγέλουν μια δραματική κατάσταση με χιλιάδε ανθρώπου μετανάστε που ζουν στο δρόμο στη Βέλικα Γκλάτουτσα και στον Μπίατς σε συνθήκες πραγματικά απαράδεκτες χωρίς ε, σωστή ε, ιατρική ε, ή νομική υποστήριξη. Και μάλιστα σύμφωνα με τον Guardian τους τελευταίους μήνες υπήρξε συστηματική χρήση βίας εκ μέρους των κροατικών αρχών στα σύνορα αυτά για να αποθήσουν τους ετούντες άσυλο στη Βοσνία. Θέλω να ρωτήσω αν είναι παρόν ο Frontex στα σύνορα αυτά και στην περίπτωση αυτή με πόσες μονάδες. Γιατί θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να ε, ελεγχθεί το τι συμβαίνει εκεί πέρα σύμφωνα με τις καταγγελίες από πολλές πηγές προερχόμενες. Το τελευταίο, θα ήθελα να καταλάβω αν τελευταία υπήρξε μείωση ε, των εκπομπών SOS στη Μεσόγειο ε, κοντά στα χωρικά είδωτα της Λιβύης. Γιατί μου είναι πιο δύσκολο να καταλάβω πώς λειτουργεί και τι κάνει η ακτοφυλακή της Λιβύης και τι γίνεται με το σεβασμό των ανθρώπων εκ μέρους της. Να τηρήσουμε αυτό το όριο των ε, δύο λεπτών, συνάδελφοι. Έχουμε και θέμα με τα χρωματικά με τα προτείνεται να καλυφθούν 10.000. Πού θα τους βάλετε στην Βαρσοβία. Τι υπολογισμό έχει γίνει για τους επαναπατρισμούς. Τι θα γίνει με την πλατφόρμα απόβασης. Και τα κράτη-μέλη έχουν σοβαρά προβλήματα με τους επαναπατρισμούς. Α, καλά που είπατε ότι η διαχείριση συνόρων δεν σημαίνει μόνο αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Κάθε ξέρω θα γίνουν αυτοί οι 10.000 της βρόντεξ, αλλά γιατί να είναι όλοι στα σύνορα. Θα μπορούσαν να βοηθήσουν και για το λαθρεμπόριο όπλων και λόγω. Πού νομίζετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε ούτω ώστε να ανασχέσετε αυτό το έγκλημα το οποίο όντω ε, αφορά, περνάει από τα σύνορά μας. Κέγγε. Ευχαριστώ. Κλόντ, ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Μια πάρα πολύ σύντομη ερώτηση. Όσον αφορά αυτούς τους ε, υπαλλήλους αξιωματικούς συνδέσμους για τους οποίους μας μιλήσατε, Πόσοι θα είναι, τύπο, πώς, πώς το βλέπετε, γιατί μην είπαμε πόσο σημαντική είναι. Όσον αφορά το ρόλο τους ε, για τη σχέση με τις τρίτες χώρες. Πώς μπορεί να βοηθήσουν, γιατί είπαμε ότι πρόκειται για κάποιον από κάποιο κράτος μέλος που δουλεύει στα πλαίσια της αντιπροσωπείας της Ένωσης σε ένα κράτος μέλος. Απαντήστε μου σε αυτό αν θέλετε. Καλά λέει ο κυρία Βερζιά τώρα. Όχι πάνω από δύο λεπτά παρακαλώ. Α, να, κάτι ξέρεις θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Είπαν όλοι ότι έχουμε όλο και λιγότερες μεταβάσεις από Λιβύη προ Ιταλία. Γιατί ο άραγε τι η Λιβύη σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, έχει μία ζώνη, τη ζώνη ΣΑΡ. Search and Rescue. Search and Rescue, έρευνα και διάσωση. Και συμμετέχουν και οι Ιταλοί, αλλά η αναγνώριση της ζώνης αυτής δεν σημαίνει ότι η χώρα είναι ασφαλής, αλλά σε αυτό το πλαίσιο, για πέστε μου, πόση σοφία, πόση ένωση παρεμβαίνει. Γιατί έχουμε κάποια στατιστικά το Σεπτέμβριο που λέει ότι από τους 10 που διαβαίνουν την Μεσόγειο, ένας φτάνει στην Μεσόγειο. Επτά παραπλωθούνται στην Λιβύη με τις γνωστές συνέπειες και οι υπόλοιποι 20% δηλαδή πνίγονται εσείς, η υπηρεσία σας δηλαδή, τι κάνετε σε σχέση και με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μάρια Κριστίν, σε ευχαριστούμε. Χώρα Φερνάντο, και εσύ να είσαι σύντομος. Διευθυντά δύο ερωτήματα. Πήγα προσωπικά και είδα στην Νότια Ελλάδα και η Ιταλία τα σημεία απόβαση αποβίβασης και εκεί ήταν παρούσα η Frontex, του είδα. Και στη χώρα μου, στη Νότια Ισπανία, Θέουτα, Μελίγια, Γιβραλτάρ κλπ. Τι γίνεται εκεί. Δεν υπάρχει συνεργασία με τα κράτη. Επίση, τι τεχνικές δυσκολίες υπάρχουν που σας εμποδίζουν να είστε αποτελεσματικοί ως Frontex. που εμποδίζουν τις συμπληρωματικές ενέργειες των κρατών μελών όσον αφορά τη φύλαξη των συνόρων και των ακτών. Ένα λεπτό, ένα λεπτό μίλησα. Όχι, δύο πρόεδρε. Καλά, καλά λέει ο δεν έχουμε καιρό. Γκόμες. Να απαντήσω για την Λιβύη. Εκτός από αυτά που σας είπαν. Ναι. Τι γίνεται με το εμπόριο θεωρήσεων διαβατηρίων στην Μάλτα για πρόσωπα που έρχονται από την Αφρική Και σε σχέση με αυτό που ο κύριος Αγγιλάρ τι γίνεται στην Μελίγια, τι γίνεται και στην Βόρεια Αφρική από πλευρά Frontex, είναι σαφές ότι οι λαθροδιακινητές κάνουν ό,τι θέλουν, αλωνίζουν. Αφήστε που έχουμε εκεί πέρα και ξύλιμα χρήματος. Τι πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εκεί, ο πρόεδρος. Κοιτάξτε, έχουμε το επόμενο θέμα. Έχουμε άλλον ένα διευθυντή του FRA. Οπότε τώρα ροκανίζουμε από το δικό σας χρόνο. Ε, και θα περάσουμε τελικά το όριο του 12.30. Αυτό είναι, είναι και θέμα των διερμηνέων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο κ. Λετζέρη. Ευχαριστώ τα αξιότιμα μέλη για τις ερωτήσεις σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Λιβύη γενικότερα. Ε, οφείλω να πω ότι ο, ο ίδιος ο Frontex δεν ασκεί εξωτερική πολιτική ή διπλωματία. Είμαστε επιχειρησιακός οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οφείλουμε να τηρούμε την εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Αυτό που μπορώ να πω πάντως είναι ότι δεν έχουμε κανένα επιτόπου στην Λιβύη. Δεν έχουμε άξιωματικού συνδέσμους ή παρουσία στην Λιβύη. Είναι δύσκολο λοιπόν για μένα να σας δώσω ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει εκεί. Αυτό που γνωρίζουμε, όσα, τα, όσα γνωρίζουμε, είναι από ανοιχτέ πηγές. Και πάντως δεν νομίζω ότι μπορώ να χαρακτηρίσω την ε, Λιβύη ως την καλύτερη χώρα του κόσμου. Και θα ήθελα βέβαια να πω επίσης ότι σε ό,τι αφορά τη ζώνη έρευνα και διάσωση που έχει ορίσει η Λιβέη, τη γνωρίζουμε, αλλά δεν μοιραζόμαστε πληροφορίε με τις λιβικές αρχές. Και αυτό είπα και στην έκθεσή μου, όταν είπα ότι υπάρχουν νέες καταστάσεις που δεν προβλέπονταν το 2014. Αυτή η νέα κατάσταση είναι ότι, για παράδειγμα, έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε εμείς εξαέρος επόπτευση και όπου θεωρούμε ότι υπάρχουν καταστάσεις ενδιαφέροντος, δηλαδή περιπτώσεις έρευνας και διάσωσης και έχουμε συμβάλει σε διασώσεις από ευρωπαϊκά μέσα, επιμένω, είτε ευρωπαϊκής χώρας μέλους, είτε του ίδιου του Frontex. και μια φορά ήταν ένα σκάφο την Ισίας, γιατί ήταν κοντά στην την Ισιακή ακτή. Και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Search and Rescue ήρθε σε ε, επαφή με, του, με τις νησιακές αρχές, αλλά η μία περίπτωση. Δεν υπάρχει πλαίσιο για ανταλλαγή πληροφοριών με γειτονικέ χώρες ή ε, συνομιλητές σε γειτονικέ χώρες. Έως τώρα δεν ανταλλάσσουν πληροφορίες με Λιβύη. Αλλάζω στα γερμανικά τώρα. Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν υπήρξαν ποτέ αποβιβάσεις από σκάφη του Frontex στην Λιβύη. Δεν έχει υπάρξει ποτέ τέτοιο πράγμα. Όταν ακούω πότε θα έχουμε την πρόθεση να επαναλάβουμε τέτοιου αποβιβάσει, δεν μπορώ να συμφωνήσω, διότι δεν υπήρξαν ποτέ. Το τονίζω. Συνεχίζω στα αγγλικά. Τα κριτήρια για την έρευνα και διάσωση και ο τρόπος που οργανώνεται η έρευνα και διάσωση στην κεντρική Μεσόγειο. Ανταλλάσσουμε πληροφορίε με χώρες μέλη της Ένωσης που βρίσκονται στην άμεση γειτονία. Αυτό σημαίνει Ιταλικές αρχές ή Μαλτέζικες αρχές έρευνας και διάσωσης. Εάν πρόκειται για κάτι το οποίο δεν είναι στα πλαίσια της θέμηδος, εάν είναι στα πλαίσια της θέμηδος, τότε το διαχειρίζονται οι Ιταλικές αρχές. Εδώ δεν έχω τίποτα ιδιαίτερο να πω. Ε, το 2017 η ερώτηση που έγινε ήταν σχετικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων έρευνα και διάσωση που διενήργησε ο Frontex. Σα τα λέω από μνήμη τώρα. Περίπου 25% όλων των ε, δράσεων έρευνα και διάσωση που έγιναν, έγιναν μάλλον από τον Frontex. 25% από τι συνολικέ δράσει Search and Rescue το 2017 αναλήφθηκαν από τον Frontex. Και αν θυμούμε καλά, μη κρατικές οργανώσεις έκαναν άλλο 25% των ε, ερευνών και διασώσεων. Ο λόγος είναι ότι η Uniformed, Σοφία, δρά στις περιοχές όπου δρούν οι NGO και αυτό είναι πολύ κοντά στην Λιβύη. Ενώ η επιχειρησιακή περιοχή του Τρίτονος είναι λίγο πιο βόρεια η επίπτωση μέτρων που αποφασίστηκαν από την Ιταλική κυβέρνηση για, τους, για τις μη κρατικές οργανώσεις. Πρόκειται για κώδικα δεοντολογίας που εγκρίθηκε στην Ιταλία το καλοκαίρι του 2017 για NGO. Και εξ όσων γνωρίζω δεν έχει υπάρξει άλλος πρόσθετος κώδικας διοντολογίας για τη συνεργασία με τις μη κρατικές οργανώσεις. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι από την, από την σκοπιά του Frontex αυτό που χρειαζόταν το 2017 ήταν βελτίωση της συνεργασίας και της οργάνωσης ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος, να μην υπάρχουν ενδείξεις δηλαδή ε, ε, εγκληματικής διείσδυσης δεν έγινε αλλά η, συλλογή δεδομένων εγκληματικών δραστηριοτήτων είναι επαγγελματική υπόθεση ε, που πρέπει να γίνεται από τους ε, ε, κατάλληλους αξιωματούχους. Μιλήσατε και για κάτι που ίσως φανεί ως διάκριση βάρος του Frontex από τη θεσμική πλευρά, από την νομοθετική πλευρά. Αυτό που εννοώ και πάλι βέβαια το πλαίσιο είναι διαφορετικό από ό,τι ήταν το 2014. Αυτό που εννοώ είναι αυτή η τριμερή συνεργασία με ΕΜΣΑ και ΕΦΚΑ. Για να δώσω ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Εάν το σκάφος τη Fishering Control Agency προβαίνει σε μία δράση, μπορεί να αποβιβάσει σε τρίτες χώρες, με πλήρη σεβασμό βέβαια, της αρχής της μία επαναπρόθεσης που σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο και εδώ είναι το παράδοξο κάποιες χώρες μέλη στην πρόσω μπορεί ε, να έχουν τον πειρασμό, να πέσουν τον πειρασμό να μην χρησιμοποιήσουν τον Frontex και να χρησιμοποιήσουν άλλους φορείς για την αποβίβαση διασωσμένων μεταναστών σε τρίτες χώρες. Αυτό λέω όταν, αυτό εννοώ μάλλον όταν μιλώ για διάκριση σε βάρος του Frontex. υπήρξε ένα είδος διακρίσεως τέτοιο. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα, η δέσμη μέτρων για τη διαλειτουργικότητα έχει τον στόχο να τα διορθώσει αυτά τα κενά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των διασωθέντων, πέρσι σε σχέση με το 2014, ο οργανισμός διέσωσε 34.000 άτομα. και φέτος 30.000. Είναι η εντολή μας από το 2016. Αυτό σημαίνει ότι όταν είμαστε παρόντες κάπου, στα εξωτερικά ναυτικά σύνορα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και τα πληρώματα μας είναι εκπαιδευμένα να παρεμβαίνουν ως φορείς δράσης έρευνα και διάσωση. ανά πάσα στιγμή. Αυτό που μπορώ να πω σχετικά με το χερσαίο Κροατία, βοσνιας Εκεί έχουμε αναπτύξει αεροσκάφος το οποίο υπερίπταται των συνόρων αυτών στον κροατικό εναέριο χώρο και μπορούμε να εντοπίζουμε ομάδες μεταναστών αλλά ορισμένες φορές και εγκληματικές δραστηριότητες. Όμως επιτόπου χερσαία δεν είμαστε ανεπτυγμένοι διότι δεν έχουν ζητήσει οι κροατικές αρχές. Τώρα, σχετικά με τον ρόλο των αξιωματικών συνδέσμων και τις μελλοντικέ επαφές ε, και σχετικά με τις βίζες. Ο ρόλος των αξιωματικών συνδέσμων είναι να διευκολύνουν τις σχέσεις με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, για παράδειγμα στην Τουρκία. Ο αξιωματικός σύνδεσμός μας έρχεται σε επαφή, διευκολύνει τις επαφές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας Έχουμε και διαφορετική συνεργασία με την Τουρκία. Ο ξεχωματικός σύνδεσμος μπορεί λοιπόν να συμβάλλει σε αυτά. Στον Νίγηρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πρόκειται για συνεργασία με τις αρχές του Νίγηρα που έχουν ευρύτερο ε, πεδίο εφαρμογής, δεν αναφέρονται μοναχά σε θέματα μετανάστευσης. Ε, προσφέρουμε και τεχνική στήριξη και επίσης με CSTP UCAP Niger, δηλαδή με την αποστολή που είναι επιτόπου στο Νίγηρα. Στα Δυτικά Βαλκάνια, επίση, η δράση μα σχετίζεται περισσότερο με την προετοιμασία τη ένταξη. Ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή, ο ρόλο μα μπορεί να είναι διαφορετικό δηλαδή. Όσον αφορά το μέλλον και τον ε, ε, φοδιασμό μας με 10.000 υπαλλήλους και πού, πώς το βλέπω αυτό, Νομίζω ότι πρέπει να δούμε το υπάρχον ε, σώμα σαν μια στρατηγική δεξαμενή για την ευρωπαϊκή ε, συνοριοφυλακή που μπορεί να καλύψει κάποια κενά στα κράτη-μέλη, ανάλογα με ε, τις ε, εκτιμήσεις. 5.000 ε, ε, συνοριοφύλακες λείπουν, δεν λέμε ακριβώς σε ποιο κράτος, αλλά υπάρχει ένα διαρθρωτικό έλλειμμα. Λείπουν 5.000 συνοριοφύλακες. Από το μισό από αυτό το υπάρχον σώμα είναι πάρα πολύ ευέλικτο και θα μπορούσε να αντιμετωπίσει εποχιακά, εποχιακά κενά που ε, υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέλη, όχι μόνο για θέματα μετανάστευση, αλλά για να λειτουργούν σωστά και τα αεροδρόμια. Επίση, πρέπει να δούμε ότι η διαχείριση των ε, συνόρων πρέπει να διευκολύνει την νόμιμη διαέλευση. Είναι απαράδεκτο ε, οι ταξιδιώτε να πρέπει να περιμένουν ώρε σε ένα αεροδρόμιο ή σε ένα χερσαίο σημείο διέλευση λόγω των προβλημάτων προβλημάτων υπάρχουν. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε και αυτό. Και σίγουρα ε, ένα μεγάλο μέρο των 10 θα μπορούσαν να καλύψουν τα εφιστάμενα κενά και θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν αν έχουν τις κατάλληλες νομικές ε, αρμοδιότητες για να υποστηρίξουν τις ε, εθνικές αρχές στις διαδικασίες επιβολής του νόμου, συλλογή στοιχείων, διαβίβαση στοιχείων φυσικά πάντοτε στα πλαίσια του Ευρωπαίου Επόπτη ε, Προστασίας των Δεδομένων με διαφάνεια και μέσα στο υπάρχον νομικό πλαίσιο. Τώρα για το τελευταίο τελευταίο ερώτημα για τη θεώρηση στη Μάλτα, το, τη Βίζα. Ε, δυστυχώς ε, ο Frontex δεν έχει καμιά αρμοδιότητα για την πολιτική ε, θεωρήσεων και εδώ πάλι διαβάζουμε κι εμείς από ανοιχτέ πηγές, ε, εκθέσεις του Κοινοβουλίου, ε, επιστολές που αποστέλλονται από θεσμικά όργανα Τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε άλλα θεσμικά όργανα ή σε άλλους οργανισμούς. Ε, Δυστυχώ δεν μπορώ να σα πω τίποτα περισσότερο γιατί ο Frontex δεν έχει καμία ανάμειξη σε τέτοιε υποθέσει. Ευχαριστώ συνάδελφοι, λέει ο πρόεδρο. Ξέρω ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα πετούσε περισσότερο διάλογο, θα μπορούσαμε να πάμε σε μεγαλύτερο βάθο και να ε, απαντήσουμε και σε κάποιε από τι απαντήσει που δόθηκαν. Αλλά δυστυχώς ε, δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε φάει χρόνο και από, την, από το επόμενο σημείο τη ημερησία διάταξη. Ε, δυστυχώς λοιπόν δεν μπορούμε να, να επεκταθούμε, πάντως θα δοθεί συνέχεια πολύ ε, σύντομα από τον Frontex. Θα ξανακούσουμε πολύ σύντομα από τον κύριο Λετζέρη. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ τον ε, εισηγητή και όλα τα μέλη. Okay, colleagues, uh, starting a... Συνάδελφοι, έχουμε αργήσει και συμπαθάτε αλλά θα πρέπει τώρα να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων γιατί έχουμε την 70η επέτειο της διακήρυξης δικαιωμάτων του ανθρώπου. Με, είναι τιμή μας που έχουμε εδώ τον Μάικλ Οφλάχερτη που είναι ο διευθυντής του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, FRA. Ήδη έχει κοπεί ένα τμήμα, έχει, έχει, έχει ένα τμήμα του χρόνου μας Οπότε θα πρέπει να δούμε και την επίγεια των δερμηνέων. Οπότε έχουμε τώρα την 70η ε, επέτειο της Οικονομικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και επίσης ε, έχουμε και το ζήτημα ε, της παρουσίας των προτάσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δράσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ. Τα θέματα επομένω εδώ είναι ευρύτατα και πολλά. Ε, γι' αυτό έχουμε εδώ τον Μάικλ, ο οποίος θα μας μίλησε και πρόκειται να μας διαφωτίσει. Αλλά κάτι σχετικό θα συζητήσουμε και σήμερα το απόγευμα. Πε μα για να δούμε και στο υπέτειο τη κομμουνική διακήρυξης, Μάικλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, όντω πρόκειται σε λίγε μέρε για την 70η επέτειο τη Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων Ανθρώπου. Και είναι η τέταρτη φορά που ε, σε αυτή την ε, δεκαετία, σε μια τέσσερα κονταετία έχουμε τέτοια επέτειο. Πρώτη φορά το 1988 ήμουν στο Πανεπιστήμιο και ενδιαφέρομαι για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και είχαμε τότε την 30η, 40η επέτειο. Από τότε όμως, θεωρείται στην δυτική τότε Ευρώπη άσχετο θέμα, τα θέμα των δικαιωμάτων. Αλλά στο Ανατολικό Μπλοκ είχαμε τις επαναστάσεις τους ξεσηκωμούς που οδήγησαν στις ανατρεπτικές εξελίξεις στην δεκαετία του 90. Επομένως, να μην ευχαριστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 88, το 98, το 98 στη Σιέρα είχαμε αυτόν τον εμφύλιο και εκεί κάναμε κάποιες εκδηλώσει των ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δύο εβδομάδες μετά οι επαναστάτες ε, ισοπαίδωσαν αυτή την έκθεση, οπότε πρόκειται για ένα αποτρόπιο πόλεμο, αλλά αυτό συμπίπτει με την ίδρυση, τη συγκρότηση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Άρα απελπισία αλλά και ευκαιρία. Το 2008 σε όλο τον κόσμο είχαμε την οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις στον άνθρωπο ακόμα είναι αισθητέ παντού. Οπότε τότε κάναμε και κάποια κριτήρια εδώ στις Βρυξέλλες όσον αφορά την υπηρεσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Χάρτη Ανθρωπίνων ε, Δικαιωμάτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση που τότε ξεκίνησε τη διαδρομή της. Άρα ευκαιρίες και σκοτεινά σημεία. Έχουμε επομένω ε, το ζήτημα των απειλών, το των σήμερα ζωντανών απειλών που συζητάει συνέχεια. Τώρα πάντως όταν συνθήκαμε στην ε, Βιέννη στο φόρουμ είχαμε 700 άτομα από όλη την Ευρώπη, πολλούς εξημών. Οπότε μπορώ να σα ευχαριστήσω που στείλατε αντιπροσωπεία στο φόρουμ εκείνο. Κύριε Κίνγκη, ήταν επικεφαλής αυτής της αποστολής, αλλά και εσείς, ε, Πρόεδρε, που ήρθατε στο φόρουμ. Οπότε σε αυτούς τους σκοτεινούς κύρους, έχουμε, έχουμε στοιχεία είναι, είναι βάσιμη η αισιοδοξία που τρέφουμε και για να δούμε τώρα τρία σημαντικά μέτωπα εκεί που όλοι μας ε, ανησυχούμε για αυτά τα μέτωπα διότι συζητήσατε πριν από λίγο για τη μετανάστευση η υπηρεσία μας επανειλημμένα έχει γνωμοδοτήσει προς εσάς για πάρα πολλά ζητήματα και για τα πιο δύσκολα οπότε μπορέσαμε να σας δώσουμε έρευνα εις βάθος σας πούμε τι ισχύει, τι μάθαμε από την ε, παρουσία μας στα κέντρα καταγραφής, στα hot spots σε Ελλάδα, Ιταλία και αλλού και μεταξύ των άλλων που μας ε, ανησυχούν είναι τα εξή για τη μετανάστευση. Πρώτα-πρώτα όσον αφορά τις συνθήκες στα ελληνικά νησιά. Γιατί έφτασε ήδη ο χειμώνα και εκεί επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, υπερπληθυσμός θα λέγαμε, στις, στους καταλυσμούς, στα στρατόπεδα υπάρχει πρόβλημα. Και σε αυτά τα πλαίσια θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ θετικά τα προγράμματα εθελούσιας κατάσταση. Υπάρχει και πρόγραμμα που συμφωνηθεί μεταξύ Ελλάδος και Πορτογαλίας. Επίσης, ανησυχούμε για την προστασία των ανηλίκων. και συζητήσαμε τα της κράτησης των ανηλίκων, κάτι το οποίο παγίως είναι απαράδεκτο και μη αποτελεσματικό. Οπότε θα πρέπει να ερευνηθεί το τι ισχύει, γιατί υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό και ότι ο ανήλικος αυτό το οποίο χρειάζεται δεν είναι το να περιοριστεί κάπου, αλλά είναι το να του δείξει κανείς κατανόηση και να το πλησιώσει Επίσης να δει τι γίνεται με τους μετανάστες οι οποίοι πνίγονται στην Μεσόγειο το 2015 είχαμε χίλιους. Ε, τέσσερις χιλιάδες. Τέσσερις σε κάθε χίλιους που νίγονται. Και, ε, και τώρα έχουμε 24. 2,4% το 18. Τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι θέμα μόνο έρευνας και διάσωσης. Είναι το πώς θα βρούμε κάποιου διάβλους νόμιμους προς την Ευρώπη και να μην ποινικοποιείται το έργο των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Τέλος, για τη μετανάστευση πρέπει να σας πω ότι έχουμε εντατικοποίηση, έχουμε αύξηση της ε, ρητορικής μίσους και των σχετικών εγκλημάτων. Αυτό στα 14 κράτη-μέλη το οποίο έχει θίξει η μετανάστευση. Οπότε, γι' αυτό και έχει σημασία ο δικός σας ρόλος για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, όποτε ανακύπτει. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την καταπολέμηση των δυσμένων διακρίσεων. Είναι σοβαρό το πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιθωριοποιούνται αυτοί που είναι διαφορετικοί από εμά, αυτοί που δεν ανήκουν στην πλειοψηφία. Επανειλημμένα το έχουμε καταγγείλει. Έχουμε και τις σχετικές ε, έρευνες της Υπηρεσίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Να, πρόσφατα έχουμε δύο τέτοιες έρευνες. Σας τις έχουμε παρουσιάσει όσον αφορά τους ε, μουσουλμάνους μετανάστες και τους τσιγκάνους Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί βλέπουμε ότι εκεί είναι πάρα πολύ έντονες οι δυσμενείς διακρίσεις και η περιθωριοποίηση. Επίσης, τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε και άλλη έρευνα. Σε μια, σε μια εβδομάδα θα έχουμε μια νέα έρευνα. Ο τίτλος της είναι «Τι συμβαίνει με τους μαύρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Το να είναι κανείς μαύρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τα λέει όλα. Και επίσης το να είναι κανείς Εβραίος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θίγει το θέμα του αντισημιτισμού στην Ένωση, στην Ευρώπη. Για να δούμε τώρα κάτι άλλο στις λεπτομέρειε του. Πρώτα-πρώτα, έχουμε την κοινότητα των ΛΟΑΔ. εκεί έχουμε στοιχεία που κατατείνουν στο ότι υπάρχουν συνεχώς παγίως δεσμενείς διακρίσεις για τη στέγαση, την παιδεία, την υγεία κλπ. Και, και, και ξέρετε, είχαμε μια 16χρονη λεσβία που σε μια εκδήλωση που γινόταν στο κοινοβούλιο που έλεγε τι έχει πάθει, ε, τι έχει υποστεί στο σχολείο της και όχι μόνο. Μπράβο που το πρόσεξατε το ζήτημα και είχατε και τη σημερινή σας ε, συζήτηση σχετικά για ε, τον κατάλογο δράσεων και θα πρέπει να σας πω ότι το 2019 η Υπηρεσία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα ξανακάνει κάποια έρευνα για τις εμπειρίες των ΛΟΑΔ στην Ευρώπη. Αλλά θα προσθέσουμε και τους μεσοφιλικούς εκεί, ε, στους υπόλοιπους ΛΟΑΔ. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε και το απρόσωπο με αναπηρία στο θέμα μας ε, απασχολεί. Έχουμε ένα εκατομμύριο χιλιάδες συμπολίτες μας που ζουν σε ιδρύματα. Θα μπορούσε να είναι πληθυσμό μια ε, μεσαία χώρα, μικρομεσαία χώρα τέλο πάντων, για του λόγου αυτού, γιατί έχουν κάποια αναπηρία. Ε, αυτό τώρα μα απασχολεί και έχουμε μια έκθεση στι 4 Δεκεμβρίου που θα δημοσιοποιήσουμε σε σχέση με το πώ μπορεί κανεί με σεβασμό να μεταχειρίζεται αυτά τα πρόσωπα και επίσης μια τελευταία παρατήρηση για τα άτομα με αναπηρία στα πλαίσια των ευρωεκλογών. Γιατί έφτασε η ώρα να προσέξουμε περισσότερο την υπόθεση τη συμμετοχής στο πολιτικό γίγνεσθε αυτών των προσώπων. Και κάτι άλλο για τις δυσμενείς διακρίσεις γενικότερο. Έχουμε πάγια δέσμευση ως υπηρεσία να υποστηρίζουμε πάσα πρωτοβουλία από τα θεσμικά όργανα ούτως ώστε να ισχύσει η οδηγία για την ίση μεταχείριση που είναι τόσο απαραίτητη. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Είναι αυτονόητο. Δεν νομίζω ότι θα διαφωνούσε κανείς από εσά ότι θα πρέπει να, οι δικαστές να εργάζονται ελεύθερα. Αυτό είναι εκ των ανούκανευ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου για αυτή την, το, τον κοινό χώρο δικαιοσύνης της Ένωσης, αλλά και για να υπάρχει μια υγιής οικονομία στην κοινωνία μας. Είναι κομβικό θέμα να λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο τα δικαστήρια. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ θετικό το ότι και αυτό το θέμα το προσέχει η Επιτροπή σας. Και θετικό του είσαστε πρωτοπόροι σε αυτή την προσπάθεια. Και πρόσφατα. Θεώρησα πάρα πολύ θετικό το ότι διατυπώσατε αυτή την πρόταση για να θωρακιστεί η πρωτοβουλία της Επιτροπής για αυτό το πρόγραμμα δικαιωμάτων και αξιών. Σας διαβεβαιώ, εμείς έχουμε στρατευτεί ως υπηρεσία και σε σχέση με το δικό σας έργο θα πρέπει να στηριχθείτε στα δεδομένα που έχουμε στην ανάλυση μας ε, στο υλικό που σας δίνουμε και αυτό θα αφορά και την προσπάθεια του χρόνου για το σύστημα των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων τα οποία ε, το οποίο θα σας ε, εξηγήσω αν θέλετε τώρα δεν φτάσουμε στο τέλος της διαδρομής πριν τα πράγματα βελτιωθούν θα γίνουν χειρότερα είμαι βέβαιος ότι τελικά θα τα καταφέρουμε ότι τελικά τα πράγματα θα βελτιωθούν γιατί ε, προσφέρουν έμπνευση οι νέοι. Σήμερα έχουν μαζευτεί κάπου εδώ, σε αυτό το κτίριο. Και νομίζω ότι θα μας βγάλουν από το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε, αλλά επίσης και βραχή πρόθεσμα Υπάρχουν ευκαιρίες, θα πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε. Να, ενδεικτικά για του χρόνου έχουμε την δεκάτη επέτειο του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό δεν μπορεί να είναι μόνο μία ε, μία ημέρα συζήτησης. Πρέπει να είναι η ευκαιρία να πάρουμε αυτό το εξαιρετικό νομικό πλαίσιο και ε, όργανο, μέσο για να του δώσουμε τη ζωή που ε, είχαν ε, υπόψη τους οι εμπνευστέ του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική ομιλία, Μάικλ. Ε, χρειαζόταν ένα χειροκρότημα, σίγουρα. Δύο πράγματα σκεφτόμουν. Πώς το καλό μπορούμε να συζητάμε την οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τον ρόλο που παίζει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, ε, μέσα σε 20 λεπτά είναι αδύνατον. Αλλά μου αρέσει αυτό που κάνεις, Μάικλ, που ε, <laughs> βγάζεις το λόγο σου ε, χωρίς να δίνεις δεκάρα για τίποτα άλλο. Είχαμε ε, αυτό το θέμα όμως στην ημερήσια διάταξη, ε, τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που γίνεται ε, κάτι όλο και πιο ασαφές στις μέρες μας και στην ομιλία σου έδωσες μερικά πολύ καλά παραδείγματα περί του τι πρόκειται. Μιλήσατε για τη Μεσόγειο, για την οριζόντια οδηγία περί μη διάκρισης και πολλά άλλα παραδείγματα ε, που είναι ένα πολύ καλό σχέδιο για μας. Και εμείς ε, έχουμε μια πολύ καλή αντιπροσωπεία στον ε, Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα με επικεφαλής Σεσίλια. Πολύ ωραία λοιπόν όλα αυτά. Οι διερμηνείς τώρα θα πρέπει να φύγουν δυστυχώς οι διερμηνείς θα μπορούσαν να μεταφράσουν μόνο την Κριστίν. Κριστίν, συνέχισε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. It is a great anniversary that we are celebrating today. But my enthusiasm for this fundamental text for human rights is mixed with my concern